καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Στο συγγνώμη σας έκανα να περιμένετε για μερικά λεπτά. Και ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Πρώτο σημείο, εγκρίση ημερησίας διάταξης. Και αν δεν έχετε άλλα σχόλια, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη χωρίς αλλαγές. Δεν βλέπω σχόλια. Ανακοινώσει του Προέδρου. Είναι συντομία. Η κοινή επιτροπή με την Επιτροπή Πολιτισμού. 13 Ιουλίου, 5η, 5 με 6.30. Το απόγευμα. Για να εξετάσουμε ένα σχέδιο έκθεση σχετικό με μια συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική για τον πολιτισμό και τις δημιουργ... τους δημιουργικούς κλάδους, τον κλάδο της δημιουργίας. 13 Ιουλίου λοιπόν. 3. Έγκριση πρακτικών. Έχετε λάβει τα πρακτικά της 16ης και 17ης Μαρτίου και 7ης Απριλίου. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια θα θεωρηθεί πως συγκρίνονται τα πρακτικά. Εγκρίνονται λοιπόν και σας ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στην ε, δημόσια ακρόαση για το πακέτο για το φυσικό αέριο, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας και καλωσορίζω τους ομιλητές μας, ευχαριστώντας τους για την παρουσία τους όλους ομιλητές των δύο πάνελ, των δύο τμήματων της συζήτησης. Εκ μέρους Επιτροπής, λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την ε, αποδοχή της πρόσκλησης να συμμετάσχετε στην ακρόασή μας. Είναι πολύ σημαντική αυτή. Κομμάτι του νομοθετικού έργου για το πακέτο μέτρων για το φυσικό αέριο της Επιτροπής μας. Ξέρετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πακέτο μέτρων. και έχει να κάνει με την ε, ενίσχυση της ιστορικής ε, ε, αγοράς ενέργειας και της ασφάλειας στην προμήθεια της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει λοιπόν να κάνει και με την ιστορική αγορά της ενέργειας και βέβαια με το πολύ στενά συνδεδεμένο θέμα της ασφάλειας στην προμήθεια της ενέργειας. Έχουμε τέσσερις προτάσεις, δύο νομοθετικές, κανονισμό ρύθμισης της προμήθειας με συγκεκριτή τον υποφερνόμενο, την απόφαση διακυβερνητικές αποφάσεις με τον κύριο Κρασνοντέψη εισηγητή και έχουμε δύο ανακοινώσει για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση αερίου με τον κύριο Γκιούρκ και την ψήξη και θέρμανση τον κύριο Γκίρεκ. Θα είναι ενδιαφέρουσα αυτή η περίοδος για την Επιτροπή μας. Ιδιαίτερα από το φυσικό αέριο, την προμήθεια, την αγορά του φυσικού αερίου, του φυσικού αερίου, για το φυσικό αέριο γενικά ως πηγή ενέργειας, με βάση βέβαια και την πρόσφατη ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι σημαντικό βέβαια αντίκτυπο στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακάλυψη η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει και στην ε, τήρηση του θεματολογίου της COP21. Όπως εξηγούσα λοιπόν έχουμε δύο ώρες στη διάθεσή μας με δύο τμήματα συζήτησης. Το καθένα ξεκινάει, το καθένα τελειώνει μάλλον με ερωταποκρίσεις. Και το πρώτο θέμα είναι πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία στην ενεργειακή ασφάλεια. Πρόκειται για το πάνελ υπαριθμό 1. Ταυτόχρονα βέβαια συζητούμε και το, τη δέσμη μέτρων για το φυσικό αέριο και παρακαλώ τους ομιλητές μας να περιοριστούν ο καθένας σε 8 λεπτά χρόνο ομιλίας. Ξέρω ότι δεν είναι πάντα εύκολο αυτό για σας που είστε ειδικοί του κλάδου δεν θα είναι εύκολο να περιοριστεί σε 8 λεπτά και οι συναδελφοί μας βέβαια πάντα δυσκολεύονται. Αλλά εκείνοι δεν θα έχουν, το, δεν θα έχουν παρά το πολύ 2 λεπτά. Οπωσδήποτε όχι 8 κατά τη συζήτηση. Ξεκινούμε πάντως αμέσως με τους τρεις ομιλητές του πρώτου πάνελ, τον κύριο Γιάννη Σκόπατς, Διευθυντή της ε, Γραμματείας της Ενεργειακής Κοινότητας της Βιέννης, πρώην μέλος του Σλοβενικού Κοινοβουλίου και πρόεδρο της Επιτροπής του Προϋπολογισμού του Εν Κοινοβουλίου, αλλά και υπουργό, πρώην Υπουργό των Οικονομικών, της, του περιβάλλοντος, της χωροταξίας, της ενέργειας της Σλοβενίας. Μεγάλο Υπουργείο. μεγάλα υπουργεία. Και πριν να αναλάβετε αυτά τα καθήκοντα που έχετε τώρα ως διευθυντής, ήσασταν Γενικός Γραμματέας της ε, Ενεργειακής Διεύθυνσης Σλοβενικής ε, Κυβέρνησης του Ενεργειακού Υπουργείου Οικονομίας. Γιάννης, έχεις το λόγο. Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Με τιμά. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι να σας μιλήσω. Και βέβαια θα ήθελα να σας πείσω για το πόσο καλές είναι κάποιες από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γιατί δεν εκπροσωπώ την Επιτροπή. Η ενεργειακή κοινότητα ως αναπόσπαστο τμήμα της Ενεργειακής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ενεργειακή Κοινότητα είναι τα συμβαλόμενα μέρη, οκτώ το όλων, με σαφή ε, άλλη λεξάρτηση και βέβαια ε, υπολογίζουμε πάρα πολύ σε αυτό το πακέτο μέτρων και θα προσπαθήσω να εξηγήσω στο δυνατόν πιο αναλυτικά τις θέσεις μας. Στην ε, Ευρώπη βλέπετε έχουμε πληθώρα προμήθειας σε φυσικό αέριο που ξεπερνά την κατανάλωση. Βλέπετε εδώ στη γραφική παράσταση την κατανάλωση και ταυτόχρονα την προέλευση της προμήθειας σε φυσικό αέριο. Μεγαλύτερη λοιπόν η όγκη προμήθεια από ε, αυτού τη κατανάλωση. Και αν μιλούμε για μέσου όρους και στατιστικές, συνήθως λέμε ότι είναι τρεις το ράδι και τρεις το ξύδι. Ε, βέβαια τα πάντα θα εξαρτηθούν από το πού ε, εντοπίζεται ο ε, υπομέτρηση καταναλωτή στην Ευρώπη. Εδώ βλέπετε στη γραφική περάσταση ότι αναμένεται να ενισχυθεί η κατανάλωση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο μέλλον με νέους ε, προμηθευτές που εμφανίζονται όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ινδονησία, η Αυστραλία και άλλοι χώρες αξιόπιστες πολύ περισσότερο από ότι Φερρυπίν η Ρωσία ως προμηθευτής ενέργειας, φυσικού αερίου και που θα επιδιώξουν ένα στο δυνατόν πιο φθηνές ή ανταγωνιστικές για να μπορέσουν να πουλήσουν το αέριο τους και στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν πληθώρα αερίου. Η επανάσταση της ε, υδρορογμάτωσης έχει εξασφαλίσει πολύ υψηλές ποσότητες. Για το μέλλον τώρα της κατανάλωσης του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Βλέπετε ποια είναι η σημασία του υγροποιημένου φυσικού αερίου που αναμένεται να ενισχυθεί. Οι εισαγωγέ από την Ρωσία αναμένεται να ε, μειωθούν, όπως άλλωστε και η ενδογενής, η εγχώρια παραγωγή, οι κατοχώρες, ε, Νορβηγία και άλλη παραγωγή που αναμένεται να μειώσουν ακόμη την παραγωγή του, Ωστόσο, μπαίνει στη, ε, στο προσκήνιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Υπάρχει μάλιστα μια τοποθέτηση της Επιτροπής με την στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, όπως την αναφέρει. Το νέο αυτό στοιχείο δηλαδή, την νέα αυτή υποδομή που κατά πάσα πιθανότητα θα ε, σώσει την Ευρώπη από οδήποτε κίνδυνο σπάνιδους ε, φυσικού αερίου στο μέλλον. Ο πίνακας πάντως βλέπετε εδώ δείχνει μια διαφορετική εικόνα. Μας δείχνει πού είναι ανταγωνιστική η προμήθεια, πιο ανταγωνιστική, ε, το πιο ανταγωνιστικό επίπεδο το βλέπετε στις πράσινες, ε, στις χώρες τον με πράσινο, ενώ αυτές που έχουν το κοκκινοπό χρώμα έχουν χαμηλή διαφοροποίηση προμήθειας, επιτοπλίστων δηλαδή εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο ή κατά κύριο λόγο από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Και εδώ είναι τα κύρια προβλήματα ως προς την ασφάλεια της Ευρώπης, στην προμήθεια φυσικού αερίου. Επομένως, όταν μιλούμε για ασφάλεια, προμήθεια σε φυσικό αέριο, κατά κύριο λόγο μιλούμε για προβλήματα που έχουν να κάνουν με την προμήθεια σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Γιατί όλοι οι άλλοι καταγραφόμενοι κίνδυνοι είναι επιτοπλίστων θεωρητικοί τουλάχιστον με τις δεδομένες συνθήκες. Επίσης εδώ στους δύο αυτούς χάρτες βλέπετε τεστ αντοχής του 2014 πραγματοποιήθηκαν ε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας ε, με τους κινδύνους σε περίπτωση διατάραξης της προμήθειας από τη Ρωσία. Από τη μια πλευρά στην αριστερή δηλαδή έχετε τη συντονισμένη προσέγγιση, δεξιά έχετε τη μη συντονισμένη προσέγγιση, προσέγγιση δηλαδή όπου η κάθε χώρα θα αντιδρά, θα αντιδρούσε ή θα λειτουργούσε, θα δραστηριοποιούνταν μόνη της. Εκεί βλέπετε ότι έχουμε χώρες σε βαθύ κόκκινο, ακόμη και σε σκούρο μπορντό, που δείχνουν ότι μπορεί να έχουν προβλήματα ως προς την προμήθεια, εάν διαταραχθεί αυτή από πλευράς Ρωσίας. Και εδώ έχουμε ένα χάρτη, ο οποίος δείχνει αγωγούς, οι οποίοι καταφτάνουν, φτάνουν στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό έδαφος. Έχουμε ένα γράφημα στα δεξιά με ένα πίνακα, ο οποίος δείχνει ε, την ε, φόρτωση των διαφορών αγωγών. κάποια από ό,τι βλέπετε έχουν χαμηλά ποσοστά φόρτωσης, φυσικού αερίου πάντα η αγωγή, ενώ όταν έχουμε να κάνουμε με τερματικά φυσικού, υγροποιημένου φυσικού αερίου, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, γιατί είναι πολύ μικρά τα ποσοστά ε, εξυπηρέτησης σε τερματικά ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου. Άρα μπορούμε να πούμε ότι για τις μείζονε υποδομές είναι επαρκής η προμήθεια με βάση τους αγωγούς αυτού σε φυσικό αέριο, αλλά προβλήματα ε, υφίστανται και αυτά έχουν να κάνουν με το ανατολικό κομμάτι του χάρτη της ε, Ευρώπης, αυτό που σας έδειξα νωρίτερα, σε σχέση με ενδεχόμενα προβλήματα στην προμήθεια φυσικού αερίου. Και μια από τι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η λεγόμενη ΣΥΣΕΚ, e συνδεσιμότητα κεντρικής ανατολικής νοτιοανατολικής Ευρώπης προσπαθεί να αποσυμφορήσει ορισμένα τμήματα των αγωγών στα πιο προβληματικά του σημεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Βλέπετε ότι κυρίως αφορά την νοτιοανατολική Ευρώπη. Και αυτό βέβαια, αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει και το ανατολικό τμήμα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποσυμφορήσει κάποιους από τους του ε, ή τους δρόμους προμήθειας του φυσικού αερίου. Βλέπετε τις κόκκινες γραμμές στη συνέχεια με τη χρηματοδότηση εν μέρη από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό πάλι με στόχο την αποσυμφόρηση των ε, διάβλων, των διόδων ε, διέλευσης του αερίου. Κομμάτι της ενεργειακής κοινότητας τώρα βλέπετε εδώ Εννέα είναι τα μέλη, οι χώρε με το κίτρινο είναι λοιπά συμβαλόμενα μέρη, δεν έχουν όλα φυσικό, δεν έχουν όλα αγορά φυσικού αερίου, τα περισσότερα όμως έχουν και βέβαια το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο από αυτά είναι η Ουκρανία. Και εδώ, κοντεύοντας να εξαντλήσω το χρόνο μου, θα ήθελα να αναφερθώ σε ε, χείριστες ή κακές πρακτικές εδώ όταν υιοθετείται ο κανονισμός για τις υποδομές για την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, διαγράφει ε, συνδέσμους μεταξύ ε, μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας. Με το άρθρο 15 του νέου κανονισμού υπάρχει μια καλή ρήτρα ανασύνδεσης, επανασύνδεσης που προσφέρει καλή νομική λύση σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα διασύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενεργειακής Κοινότητας, Ενεργειακής Ένωσης θα πω. Ε, και πιστεύω ότι αυτό το άρθρο 15 εξασφαλίζει καλύτερη ε, διαχείριση, διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πανευρωπαϊκό χώρο. Εμείς ως κοινότητα ενεργειακή προτείναμε να υπάρχει γενικώ μια ρήτρα επανασύνδεσης στην συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα. Δεν ξέρουμε όμω αν κάτι τέτοιο θα υιοθετηθεί. Πρόκειται για συνθήκη τελευταία ανάλυση και θα χρειαστούν και άλλε δράσει για να καλυφθεί αυτό το νομικό κενό, το νομοθετικό κενό. Δεν μπορώ όμω να επεκταθώ περισσότερο λόγω λήψη χρόνου. Εδώ βλέπετε τι χώρε οι οποίε θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τα ε, διασυνοριακά τους προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή περιφέρεια της ενεργειακής κοινότητας και ε, κάποιες άλλες προτάσεις που έχουμε, αλλά δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο. Όπως έλεγα για να συνοψίσω υπέρ του άρθρου 15 με το switch on clause, τη ρήτρα επανασύνδεσης, και ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθεί αυτό το μέτρο σαν μια γενική ε, λύση σε ε, κανονισμούς, σε άλλες διατάξεις, έτσι ώστε ο πανευρωπαϊκός χώρος και η εσωτερική αγορά ενέργειας να λειτουργήσουν απρόσκοπτα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Γιάννη Σκόπατς. Να προχωρήσουμε λοιπόν και έχουμε τώρα τον δεύτερο ομιλητή. Πρόκειται για την κυρία Μανών Ντιφούρ, η οποία είναι επικεφαλής της ε, ε, του γραφείου της ε, E3G ε, στις Βρυξέλλες. Αλλά πριν καταλάβει τη θέση αυτή, η κυρία Ντιφούρ εργάστηκε για την New Energy Finance της Bloomberg στο Λονδίνο και στην Νέα Υόρκη. Είχατε μία πολύ ισχυρή θέση εκεί γιατί έχετε ασχοληθεί με την συνολική αγορά άνθρακα ε, και με τις ευρωπαϊκές αγορές ε, ενέργειας ε, και έχετε συμμετάσχει στην διαρκή ανάλυση αυτών των αγορών. Επίσης έχετε εργαστεί και έχετε ασχοληθεί με την, ε, με τον σχεδιασμό ε, τέτοιων ε, καταστάσεων αλλά και προσωμιώσεων οι οποίες σε στόχο έχουν να βοηθήσουν την καλύτερη κατανόηση των τεκτενομένων και να βοηθήσουν όσους πρέπει να λάβουν σημαντικές αποφάσεις στις αποφάσεις αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ είναι μεγάλη χαρά που μπορώ να μιλήσω σήμερα εδώ για αυτό το σημαντικό θέμα. Πρέπει να σας πω ότι η E3G είναι ένας ε, κοινοφελής οργανισμός ο οποίος ε, ασχολείται ε, με θέματα άνθρακα και εκπομπών κτλ. Για να καταλάβετε την τοποθέτησή μου το, είναι σημαντικό να πούμε ότι η ασφάλεια της, του εφοδιασμού είναι σημαντική αυτή τη στιγμή, πράγμα που είχαμε να το δούμε ε, πολλά ε, χρόνια. Ε, πλέον έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών και πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί και από μόνο του σημαντική προστιθέμενη αξία. Ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα τελευταία χρόνια ε, είδαμε σημαντική μείωση και ταχύτατη μάλιστα μείωση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ε, και έχουμε δει επίσης και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ε, ε, καινούριες λύσεις, καλύτερες, ευφιέστερες μέσω των ευφυών διακοπτών και κέντρων κτλ. Τώρα ξεκινάει μια νέα φάση στην ενεργειακή ε, ολοκλήρωση ε, βεβαίως ε, και μέσω της διαμεθοριακής συνεργασίας αλλά εμείς θέλουμε πλέον να δούμε καλύτερη ολοκλήρωση και ανάμεσα στις υποδομές αερίου και ηλεκτρικού. Όλα αυτά συνδυασμένα με την προστασία του περιβάλλοντος και τους νέους περιβαλλοντικούς κλιματικούς στόχους. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω βλέποντας λίγο, μελετώντας το γενικότερο ε, πλαίσιο και μετά θα δούμε και κάποια επιπλέον βήματα που μπορούν ε, να ληφθούν. Το πρώτο είναι ότι για να ε, μελετήσουμε την αντοχή του συστήματος είναι ότι ζητήσαμε να μελετηθεί η αντοχή των δικτύων ε, ε, παροχής ε, και οι περιπτώσεις διακοπής της παροχής τα αποτελέσματα ε, στα οποία καταλήξαμε είναι ιδιαίτερα ανακουφιστικά. Ε, δηλαδή ε, βρήκαμε ότι το σύστημα και η υποδομή είναι εξαιρετικά ανθεκτική σε μεγάλες, σε έντονες περιπτώσεις, σε έντονα προβλήματα και διακοπή της παροχής. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έχουν επίσης αυξηθεί αυξηθεί τέσσερις φορές οι υποδομές οι οποίες υποβοηθούν ε, στο αποτέλεσμα αυτό. Ταυτόχρονα έχει μειωθεί σχεδόν στο 50% το κόστος μεταφοράς. Πέρα από την σημαντική αντοχή βλέπουμε και καλύτερο προγραμματισμό ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και όσον αφορά την μεταφορά και όσον αφορά τις εισαγωγές του αερίου. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι η ενεργειακή πολιτική ε, μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιες προκλήσεις. Διαπιστώνουμε ότι οι υποδομές ακολουθούν ένα σενάριο αύξησης ε, της ζήτησης. Εμείς πιστεύουμε ότι το 2010 αυξήθηκε, έφτασε στο, ε, στο πιο ψηλό ε, σημείο η ζήτηση ε, και τώρα έχει αρχίσει και πέφτει. Το δεύτερο στοιχείο ε, είναι ότι ε, και από τους διαχειριστές των δικτύων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την βιομηχανία υπάρχει, υπάρχουν σαφή αιτήματα έτσι ώστε να μελετηθεί σωστά η, προσφο... η ζήτηση του αερίου για τα επόμενα χρόνια και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει από το 2014. Εάν δούμε κάποια σενάρια ε, βάσει των οποίων καλύπτονται οι στόχοι οι κλιματικοί και ενεργειακοί για το 2030, τότε θα μειωθούν ε, οι εισαγωγές ε, αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε μετά από το 30 και μέχρι το 2050 ε, και αν κρατηθούμε σε αυτό το 2% της ε, θερμοκρασίας, τότε θα έχω, και εάν κρατήσουμε τις αρχές για οικονομία με, μηδενικό, με μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, τότε θα έχουμε όλο και λιγότερη χρήση αυτών των μορφών ενέργειας. Ε, βεβαίως εδώ στη συγκεκριμένη δέσμη δεν μπορούν να καλυφθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Ε, αλλά ε, μια και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ε, η, η ζωή τέτοιων εγκαταστάσεων είναι εξαιρετικά και ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικά μακρόπνος και ξεπερνάει και την 20 ετία, οπωσδήποτε θα πρέπει να, έχουμε, να ξεκινήσουμε από τώρα έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτήν την οικονομία μηδενικών εκπομπών. Η επιλογές ε, βεβαίως οι οποίες ε, ε, βρίσκονται μπροστά μας είναι σημαντικές γιατί τα ερωτήματα τα οποία τίθενται είναι από τη μία εάν σπαταλούμε χρήματα χωρίς λόγο και από την άλλη εάν δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους περιβαλλοντικούς κλιματικούς στόχους εάν θέλουμε ε, πραγματικά να φτάσουμε σε πιο ευφυείς υποδομές ε, ε, με ταυτόχρονη ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια βήματα τα οποία συμπεριλαμβάνουν κάποιους στόχους που θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται ε, οι υπόψη. Συμπεριλαμβάνονται ε, οι κλιματικοί στόχοι, ε, η μελέτη και επιβεβαίωση των μακροπρόθεσμων στόχων βιωσιμότητας κλπ. Εγώ θα ήθελα εδώ να επικεντρωθώ σε δύο στοιχεία κυρίως Βεβαίως η αποτελεσματική χρήση της ζήτησης ενέργειας είναι ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος έτσι ώστε ε, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και έτσι ώστε να ε, γίνει μια σωστή αξιολόγηση των ε, προτινόμενων πολιτικών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια μέσα από προληπτικά προγράμματα κλπ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε κατά την έννοια αυτή ε, μας δίνει κάποια ε, καλά παραδείγματα ε, μέσα από κινήσεις όπως ας πούμε η υποχρέωση των παρόχων και η υποχρέωση και των διαχειριστών δικτύων να συνεργάζονται μεταξύ τους. Αυτή άλλωστε η προσέγγιση επιτρέπει μεγάλες εξοικονομήσεις όταν μιλάμε για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η, ε, ολοκληρωμένη, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός των υποδομών. Δηλαδή δεν θα πρέπει να δούμε μονάχα κατά τη φάση του σχεδιασμού ε, το φυσικό αέριο, αλλά θα πρέπει ε, να δούμε την γενικότερη συνεργασία. Μπορεί κάποιοι, μπορεί κάποιοι πάροχοι να γνωρίζουν καλύτερα το αέριο, άλλοι να γνωρίζουν καλύτερα την ηλεκτρική ενέργεια. Θα πρέπει επομένως να υπάρχει καλύτερη ολοκλήρωση των συστημάτων έτσι ώστε ε, να ε, χρειάζεται όλο και λιγότερη επένδυση όσον αφορά αυτή καθεαυτή την υποδομή για το φυσικό ε, αέριο. Και βεβαίως ο κανονισμός για την ενεργειακή ασφάλεια και την, της προμήθεια δηλαδή της ενέργειας είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή εδώ βρισκόμαστε σε μια νέα φάση, ένα νέο βήμα προς την ευρωπαϊκή ε, ολοκλήρωση. Έχει ήδη ξεκινήσει τα τελευταία δέκα χρόνια, αλλά τώρα ε, προχωράει με ταχύτητα και ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Όλοι οι ομιλητές θα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε ερωτήσεις έτσι ώστε να ολοκληρώσετε τη βασική σας ομιλία. Τώρα έχουμε τον τρίτο ομιλητή, τον Άντριου Βόκερ, που είναι αντιπρόεδρος της στρατηγικής Σενιέρ Energy. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία του, διότι η Σενιέρ Energy θα ήθελε να προωθήσει τις εξαγωγές από τη ΣΥΠΑ στην Ευρώπη και αυτό είναι άκρος ενδιαφέρον ε, για εμάς. Εγώ βρέθηκα πέρσι στην Ουάσιγκτον όπου συνεδρίασε η Ήτρε και συζητήσαμε το θέμα με τους γερουσιαστές και με τους επιχειρηματίες πριν από την TTIP. Θα θέλαμε λοιπόν να τα οργανώσουμε όλα πριν από τη συμφωνία TTIP. Όπως ξέρετε λοιπόν, ε, ο κύριος Walker ασχολείται με το σκέλος ε, του μάρκετινγκ της ε, Σενιέρ. Πριν ήσασταν αντιπρόεδρος της Global LNG και, και είχατε συμμετάσχει και στην κοινοπραξία BG. Και εργαστήκατε ε, στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου, στον Ατλαντικό, στην Τρινιτάντ και στο Τομπάκο, καθώς και στην Αίγυπτο. Και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που καλέσατε την Σενίερ για να σχολιάσει όπως είπατε, ε, η Σενιέρ είναι μία αμερικανική εταιρεία που ασχολείται με εξαγωγές. Γι' αυτό θα μιλήσω για τις εξαγωγές των ΙΠΑ και θα σας μιλήσω για τις ε, τελευταίες εξελίξεις για να δούμε τι επιπτώσεις θα υπάρχουν και στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα ήθελα να σας επισύρω την ε, προσοχή στο ε, θέμα αυτό. Έχετε την έκθεση, μπορείτε να την δείτε. Και όπως είπε και ο πρόεδρος, η Σενιέρ εξάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο μετά από έναν προγραμματισμό. Έχουμε μπει στις εξαγωγές του ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου από 48 πολιτείες, ε, τον είπα. Εδώ βλέπετε, ότι είχαμε, βλέπετε πώς έχει η εγκατάσταση. Υπάρχουν πέντε τέτοιες εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή στις ΙΠΑ. Ε, στις 24 Φεβρουαρίου 2016 έγινε και η πρώτη ε, φόρτωση. Βλέπετε το Asia ε, Vision που διαπλέει τον ποτιμό Σαμπίν για να προβεί στις εξαγωγές έχουμε εννέα φορτώσεις έκτοτε και φτάσαμε σε αγορές στη Νότια Αμερική, Μέση Ανατολή, Ασία και το έβδομο φορτίο ήρθε στην Ευρώπη, πρόσφατα δηλαδή στην Πορτογαλία. Θα ήθελα να σας δώσω μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έδωσε ο κύριος Κόπατς. Βλέπετε ότι υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα στις ΗΠΑ και έτσι θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στο παγκόσμιο μείγμα υγροποιημένου φυσικού αερίου. Θα φτάσουμε σε 6 εκατομμύρια τόνους, αυτή θα είναι η παραγωγική μας ικανότητα στο παγκόσμιο μείγμα και έτσι είπα θα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένη φυσικού αερίου μέχρι το 2020 και πιστεύουμε ότι θα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μέχρι το 2025. Αυτές οι εξαγωγές έχουν ε, σοβαρούς αντικτύπους στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, όχι μόνο λόγω μεγέθους, και, αλλά και χάρη στο γεγονότο, του γεγονότος ότι εμείς είμαστε ένας ανταγωνιστικός ε, εξαγωγέας ως προς το κόστος. Έχουμε κοιτάσματα με χαμηλό κόστος. Εδώ βλέπετε το γράφημα, βλέπετε ότι υπάρχουν 800 TCF φυσικού αερίου με κόστος 3 δολάρια. Μπορούμε να φτάσουμε δηλαδή σε 800.000 κυβικά μέτρα και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Δεξιά βλέπετε ότι υπάρχει χαμηλό κόστος ε, δημιουργίας και οικοδόμησης ε, μονάδων, δηλαδή 800 δολάρια ανά τόνο, Άρα πολύ χαμηλότερο κόστος σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Είμαστε ανταγωνιστικοί ως προς το κόστος προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και με βάση τις αρχές του ελευθέρου εμπορίου θα πρέπει να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο εξαγωγών ανάλογα με τον προορισμό και τον όγκο εξαγωγών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχουν μεγάλα ευεργετήματα για την παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτά τα ευεργετήματα στρέφονται και προς την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένας βασικός αγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τα ευεργετήματα, την πλευρά αριστερά του γραφήματος. Θεωρούμε ότι υπάρχει ε, μία εξέλιξη ευρείας κλίμακας σε σχέση με τις ε, μονάδες εξαγωγής και όπως είπαμε η Αυστραλία βρίσκεται σχετικά μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κατάρ θα μπορούσε να στραφεί στην Ασία ή στον Ατλαντικό. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει ευέλικτα, ε, ε, ευέλικτους όγκους και αξίες έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά των αγορών. Η TTIP και οι διατλαντικές σχέσεις θα ακολουθήσουν αυτό το σχήμα εξαγωγών των ΙΠΑ ε, προς την Ευρώπη και πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές. Κάτι το οποίο δεν θα ίσχυε διαφορετικά. Το φυσικό αέριο φυσικά έχει πολύ χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με άλλους υδρογονάνθρακες και έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους στόχους της COP21. Επίσης, οι εισαγωγές θα, δημιουργήσουν, θα χρησιμοποιήσουμε συγχωρείτε, τις υποδομές που προϋπάρχουν. Εμείς έχουμε μεγάλη υποδομή που χρησιμοποιείται κατά 25% μόνο για πέρσι τουλάχιστον. Συμφωνούμε λοιπόν με τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ήτρε σε σχέση με τα ευεργετήματα της χρήσης και εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Όπως είπε και ο κύριος Κόπατς, χρειάζεται περισσότερη εργασία έτσι ώστε τα ευεργετήματα του υγροποιημένου φυσικού αερίου να φτάσουν σε κάθε πολίτη. Ιδιαίτερα στη Βαλτική, Νοτιοανατολική και Νοτιολική Ευρώπη, όπου δεν υπάρχουν ε, κατάλληλες υποδομές πάντα, θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προβλέψουμε μία στρατηγική υποδομή έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι δικαιούχοι σε αυτές τις περιοχές ως προς τις ε, εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Χρειάζεται λοιπόν η σωστή υποδομή. Θα πρέπει να υπάρχει διασυνδεσιμότητα με την εσωτερική αγορά και αυτό μέσα και στα πλαίσια των δασμολογικών περιορισμών. Για να συνοψίσω, οι ΙΠΑ έχουν, έχουν προβεί σε μεγάλες εξαγωγές. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν υψηλές ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην παγκόσμια αγορά. Έχει αλλάξει το παγκόσμιο πλαίσιο και υπάρχουν ευεργετήματα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ενεργειακή ασφάλεια ε, ευελιξία και αξιοπιστία της ε, αγοράς της ενέργειας. Εμείς τασόμαστε υπέρ της, ε, του ηγετικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής σας για να ανταποκριθείτε στην ολοένα και αναπτυσσόμενη αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου για να ολοκληρωθεί η εργασία και για να υπάρχουν αυτά τα ευεργετήματα να επεκταθούν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Τελειώνω λοιπόν υπερβαίνοντας το χρόνο μόνο κατά 49 δευτερόλεπτα και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Θα αρχίσουμε τώρα ερωτήσεις και απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα ε, το ΕΛΚΑ, εξ ονόματος μάλλον του ΕΛΚ, ο Κάρετς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα με την κυρία Ντιουφούρ συγκεκριμένα, ίσως να θέλουν να σχολιάσουν και οι άλλοι ομιλητέ μας. Να ρωτήσω σε σχέση με την ανθεκτικότητα των υποδομών φυσικού αερίου της Ευρώπης. Είπατε ότι με πολύ ψυχρό καιρό δεν υπάρχουν ε, διαταραχές σε σχέση με την προμήθεια από την Αρβηγία και άλλες βόρειες περιοχές, αλλά διαφοροποιήστε προς την ε, νοτιοανατολική Ευρώπη που θα μπορούσε λέτε, να κινδυνεύει σημαντικά. Ε, θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε περισσότερα για την ανθεκτικότητα του δικτύου μας στο φυσικό αέριο. Τι θα σημαίνει μια τέτοια διαταραχή στην προμήθεια. Και ίσως και οι άλλοι μιλητές θέλουν να σχολιάσουν ποια είναι τα πιο σοβαρά ε, προβλήματα συμφόρησης στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Υπάρχουν τερματικά, πολλά από αυτά δεν αξιοποιούνται επαρκώς, αλλά σημεία συμφόρηση έχουμε φερειπίν από τη Γαλλία ε, προς την Γερμανία. Και εάν υλοποιηθεί το έργο Nord Stream 2, μπορείτε να μας κάνετε μια πρόβλεψη για το πώς θα φτάνουν αυτές οι προμήθειες φυσικού αερίου μέχρι την νοτιοανατολική Ευρώπη. Εάν βγει από το χάρτη η Ουκρανία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το Nord Stream 2 θα βγάλει εκτό εκτός παιδιάς την Ουκρανία. Και έτσι θα υπάρχει αυτό το ζήτημα σε σχέση με τις πιθανές σοβαρές διαταραχές. Ευχαριστώ κυρία Κρυφίν, Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Ιδιαίτερος χαίρομαι για το γεγονός ότι κάνετε μια προσέγγιση ολιστική γενική και μας δίνετε ενδείξει ότι πρέπει να κάνουμε. Ασφάλεια λοιπόν στην προμήθεια, ανθεκτικότητα και ένα πιο αηφόρο ενεργειακό μείγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαρτάται από εξωτερικούς προμηθευτές και ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο με 50% εισαγόμενο φυσικό αέριο, με μειούμενη από 50,1 εκατομμύρια τόνου το 2010 στους 32 εκατομμύρια τόνου το 2013 η παραγωγή του φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της σημαντική υποβάθμιση των αποθεμάτων, των κοιτασμάτων τη Βορειάς Θάλασσας. Έτσι λοιπόν χρειάζεται οπωσδήποτε να ενισχυθεί η συνεργασία και η ελεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και ένα ε, σαφές ε, σχέδιο συνεργασίας. Δεν μπορεί κανείς απομονωμένος και μεμονωμένος να δώσει λύσεις και βέβαια θα σας ξαφνιάσω να σας πω ότι πρέπει να παραμείνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο και να διαδραματίσει το ρόλο του μέσα σε αυτήν σχέδια κατεπίγουσας ανάγκης σχέση με το φυσικό αέριο ασφαλώς χρειάζεται να υπάρχουν όπως άλλωστε προτείνει και το όραμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας και επίσης Πρόεδρε όταν αξιολογούμε την ασφάλεια προμήθειας πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση σχέση με την Ενεργειακή Ένωση και για τις ανανεώσιμε πηγές και για την αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας και βέβαια όταν μιλούμε για ασφάλεια ενέργειας πρέπει ταυτόχρονα θα συμπληρώσω να μιλούμε και για τιμές ενεργειακών προϊόντων για τον οικοκυριό και την βιομηχανία. 50 εκατομμύρια πολιτών επηρεάζονται καθώς βρίσκονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα σε ενεργειακή ένδυα. Ευχαριστώ κύριο Χένκελ, ECR. Τρεις σύντομες και συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον κύριο Βόκερ πρώτα. αναφερθήκατε στην φθήνουσα προμηθεία στην Ευρώπη και θέλω να ρωτήσω πρόκειται πράγματι για προμήθεια ή για απουσία ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πόρων φυσικού αερίου. Δεύτερον προς την κυρία Τιφούρ. Μια ερώτηση που έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που ήδη βέβαια τονίστηκε. Έχω όμως μια συμπληρωματική ερώτηση. Κάποιες από τις χώρες αυτές έχουν και εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας με εξάρτηση 100% από πυρηνικό καύσιμο ρωσικό. Η ανθεκτικότητα αυτή λοιπόν δεν μπορεί να λάβει υπόψη και το γεγονό ότι αν σταματήσει η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία θα σταματήσει η Ρωσία ταυτόχρονα και να προμηθεύει τι χώρε αυτέ σε πυρηνικό καύσιμο. Και για τον κύριο Κόπατς επίσης μια ερώτηση για τον Nord Stream 2. Θεωρούσα έκαθαν ότι δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να γίνει αυτός ο αγώγος για διάφορους λόγους. Μια όμως και υπάρχει τόση πληθώρα προμήθειας φυσικού αέριο. Τι τον θέλουμε. Σας ευχαριστώ. Άλλη κυρία Άντσετ. Κάποιες ερωτήσεις θέλω να κάνω σε σχέση με το πιθανό σενάριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με ευρεία ε, ή διευρυμένη τέλο πάντων ε, προμήθεια ε, φυσικού αερίου που ενδεχομένως θα διακόψει το δρόμο προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί όντως βλέπουμε ότι έχουν πλέον, υπάρχουν πλέον κοιτάσματα τα οποία έχουν ανακαλυφθεί. Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάσχεση της πορείας ε, των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα, οδηγήσει, θα οδηγούσε ας πούμε, σε συνέχιση της χρήσης των ε, ορυκτών καυσίμων. Δεύτερο, όσον αφορά το σχιστολιτικό αέριο και την υδρορυγμάτωση. Ακούσαμε κάποιες νέες ιδέες της κυρίας Εγκολέν Ρουαγιάλ στη Γαλλία, η οποία αναφέρει ότι μελετά ακόμα και το ενδεχόμενο νομικών ε, μέτρων ε, έτσι ώστε να απαγορεύσει ε, την εισαγωγή φυσικού αερίου που θα μπορούσε να είχε παραχθεί με τέτοιες διαδικασίες γιατί είναι λογικό ότι εάν απαγορεύεται η ορυθροκρημάτωση στη Γαλλία, είναι λογικό, λέω, να απαγορευθεί οποιοδήποτε αέριο έχει παραχθεί με τέτοια μέθοδο εκτός ε, των ε, ε, συνόρων. Και επομένως τίθενται κάποιοι περιορισμοί σε εισαγωγικές εταιρείε. Ρωτώ λοιπόν, υπάρχει η δυνατότητα στην Ευρώπη να μελετήσουμε γενικά το θέμα νομικών προσκομμάτων ε, ε, που θα τεθούν ε, στην εισαγωγή αερίου που θα έχει εξαχθεί με τέτοιου είδους μεθόδους. Επίσης, είναι δυνατόν να μελετηθούν περισσότερο οι δυνατότητες παύσης της, των εκπομπών μεθανίου, γιατί ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικά μολυντικές. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριο Τούρμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις για την κυρία Ντιφούρ. Δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά, αλλά ε, οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες μας λέτε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, όλες έχουν μειωτική τάση και η μόνη χώρα η οποία έχει περισσότερο γκάς είναι ε, η Βουλγαρία, ένα BCM και η Πολωνία. Στην ουσία δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πλέον ένα περιβάλλον όπου ε, θα αυξηθεί ας πούμε, η παραγωγή αερίου, αλλά ο γείτονά σα ε, λέει ότι μέχρι το 2018 ε, θα έχουμε 50 BTM παραπάνω. Επιπλέον. Γιατί βεβαίω καταλαβαίνετε ότι με 50 BCM επιπλέον οπωσδήποτε θα είχε πολύ αυξητική τάση η ευρωπαϊκή αγορά. Εάν κατάλαβα καλά τις αναλύσεις σας, ε, όσον αφορά κυρίως ε, την ε, πάυση παροχής, την διακοπή παροχής, λέμε ότι καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα εάν παραμείνουμε με την υποδομή που έχουμε, ενώ θα δημιουργήσουμε προβλήματα εάν χτίσουμε νέες υποδομές. Στο τέλος λοιπόν και έχοντας ακούσει όλα αυτά, τα αντι, αντιφατικά πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν είναι κουταμάρα λοιπόν από τη στιγμή που έχουμε ένα σύστημα που είναι καλό να θέλουμε να προσθέσουμε κάτι στο σύστημα το οποίο τελικά θα το ε, κάνει χειρότερο. Εδώ δεν μιλάμε για γεωπολιτικά, μιλάμε μόνο για λογική του συστήματος που αφορά το, το αέριο. Τέλος. Τον κύριο Σέσνερ. Μάλλον όχι, τον κύριο Walker δηλαδή, τη Σενιέρ. Τον είπα κύριο Σενιέρ, δεν είναι σωστό. Ε, εσείς λέτε ότι ε, έχετε έτοιμα τα φορτία σας, έχετε έτοιμα τα φορτηγά πλοία για να το μεταφέρουν, έχετε την δυνατότητα να δώσετε αέριο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τέλος όμως είδα μια ενδιαφέρουσα διαφάνεια Αναφερθήκατε σε χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του ε, ε, άνθρακα, αλλά δεν αναφέρεστε σε μείωση των ε, εκπομπών που επηρεάζουν το κλίμα γενικότερα. Κλιματικές λοιπόν εκπομπές του, της, της δικιάς σας παραγωγής σε σχέση ε, με τις ε, υπόλοιπες ε, παραγωγές γιατί καταλαβαίνετε ότι οι κλιματικές ότι οι εκπομπές που επηρεάζουν το κλίμα είναι πολλές. Η κυρία Λόμπες Μπερβέχο, θα τα πω ισπανικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εισηγητές. Θα ήθελα κυρίως να αναφερθώ στο φυσικό υγροποιημένο αέριο το οποίο κατά την άποψή μου αποτελεί ε, τον κύριο πυλώνα του, της ε, δέσμης του πακέτου ε, για το αέριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί ε, η Ισπανία αποτέλεσε πραγματικά ε, μια χώρα η οποία ήταν πρόδρομος στην χρήση αυτού του αερίου. Και πιστεύουμε ότι το θέμα της αποθήκευσης και της χρήσης του υγροποιημένου αερίου είναι πολύ σημαντικό. Πολλά από τα εργοστάσια όμως τα οποία θα έπρεπε ε, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μορφή ενέργειας για να ε, παράξουν ε, ηλεκτρική ενέργεια είναι κλειστά. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι υπάρχουν υποψίες παράνομων πληρωμών και επιδοτήσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η βάση του προγράμματος της ενεργειακής μεταβίβασης της Ευρωπαϊκής λέω ότι θα πρέπει να είναι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ρωτώ λοιπόν στα πλαίσια αυτή τη μετάβαση, τη ενεργειακή μετάβαση, ε, τι ρόλο μπορεί να παίξει το υγροποιημένο αέριο και τι ρόλο μπορούν και πρέπει να παίξουν οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Γιατί διαφορετικά μπορεί να έχουμε προβλήματα σαν αυτά που αντιμετωπίζουμε στην Ισπανία. Πιστεύω ότι η παρουσίαση από την πλευρά τη 3 g ήταν αρκετά σαφής. Ε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πριν ξεκινήσουμε προγράμματα τα οποία μπορεί να έχουν ε, πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο ε, περιβάλλον ή που μπορεί να περιέχουν στοιχεία τα οποία αντιτίθενται στην, στις, στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε πολλά παραδείγματα δυστυχώς στην Ισπανία, Καστόρκα, Στιχάνα κτλ. που έχουμε σημαντικά προβλήματα προβλήματα. Απ' την άλλη πλευρά και τελειώνω, ε, έχουμε στο Κατάρ αλλά και σε άλλες περιπτώσεις ε, παραγωγή αερίου σχιστολιθικού μέσα από μεθόδους οι οποίες δεν είναι δυνατές και ε, απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Α, ζητάτε το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Uh, Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω για τη Γαλλία. Ε, αυτή η Γαλλία του Σαρντεγκόλ, του Πομπιντού, ακόμα και του Σαρκοζή δεν έζησε σε κομμουνιστικά καθεστώτα και δεν έχει όμως και ε, σχιστολιθικό ε, αέριο. Δηλαδή ε, τελείως διαφορετικό, τελείως διαφορετικό πολιτικό σύστημα αλλά με μεγάλη δυνατότητα ανταλλαγών εμπορικών κτλ. Έχουμε στην Ουκρανία τώρα ένα πραξικόπημα το οποίο προκαλεί εξωτερικά, έξω από τη χώρα, ανασφάλεια όσον αφορά την ενεργειακή ε, ε, ασφάλεια και την παροχή ε, ενέργειας. Και τώρα έχουμε μια κατάσταση όπου το αέριο θα έρχεται από, την Ευρω... από, το... από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε τα αστεία, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί ε, και τώρα θα διασφαλιστεί λοιπόν αυτή η ενεργειακή ασφάλεια από τι ε, Ηνωμένε Πολιτείε τη στιγμή που μέχρι τώρα μα το διασφάλιζε την ασφάλεια αυτή η Ρωσία. Α είμαστε σοβαροί. Γιατί ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε, γιατί μπορούμε να δεχτούμε ή όχι το φυσικό αέριο που έχει παραχθεί με υδρορυγμάτωση από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Μέχρι τώρα, μέχρι τώρα δεν λαμβάνουμε καθόλου υπόψη τα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την υγροποίηση του αερίου και ένα σωρό άλλε μεθόδους που μας επιβάλλονται. Α είμαστε σοβαροί. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αν αύριο η Ρωσία δεν μας δώσει ε, αέριο, πόσοι τερματική σταθμοί πόσα πλοία, πόσες εγκαταστάσεις θα πρέπει να δημιουργηθούν έτσι ώστε ε, να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια. Όλα αυτά λοιπόν είναι ψέματα και απατηλά στοιχεία ε, για να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις τι οποίες καθόλου δεν χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν λοιπόν ερωτήσεις προς τους πάνελιστ. Ε, κύριε Κόπατς, Οκτώ χώρες παροχής ε, ενέργειας θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην Ένωση του τομέα της ενέργειας εάν εφαρμόσουν όλους τους κανονισμούς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο έχουν προχωρήσει. Προς την ε, κυρία Ντιφούρ, η ερώτηση είναι η εξής. Ε, θα δώσουμε προτεραιότητα ε, στο λογισμικό, στο software έναντι του πυρήνα, του hardcore. Μπορείτε να μας πείτε ε, περισσότερα. Και προς τον κύριο Άντριου Βόκερ, τον αντιπρόεδρο της ΣΕΝΙΕΡ, ως προς την σύγκριση των τιμών ενέργειας, είπα Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την ε, παροχή φυσικού αερίου από αγωγούς. Μιλάμε λοιπόν για την Αλγερία, για την Ορβηγία και την Ρωσία. Από τη Μέση Ανατολή, από τις ΗΠΑ και μιλάμε για την παροχή ε, ενέργειας μέσω αεραγωγών. Ε, μπορούμε να αρχίσουμε με τις απαντήσεις. Ο κύριος Κόπατς. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά, κύριε Μπούζεκ. Υπήρχαν ε, δύο ερωτήσεις προς εμένα. Η τελευταία. Κατά πόσο τα συμβαλόμενα μέρη έχουν ικανοποιήσει τις ανάγκες του τρίτου πακέτου ενέργειας. Νομίζω ότι η Ουκρανία ε, κατάφερε πλήρως ε, να μεταφέρει το ενεργειακό πακέτο εκτός από τον διαχωρισμό, το unbundling σε σχέση με τους ε, επιχειρηματικούς φορείς. Η διαδικασία είναι σχετικά επαχθής, υπάρχει ένας οδικός χάρτης για να εφαρμοστεί φέτος, ίσως το αργότερο του χρόνου. Έχει προχωρήσει όμως πάρα πολύ και ταχύτερα από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σερβία επίσης έχει μεταφέρει το νομοθετικό πλαίσιο, δεν το έχει όμως εφαρμόσει. Επίσης η Βοσνία δεν έχει μεταφέρει ακόμα το τρίτο ενεργειακό πακέτο, ούτε και η Φύρομ. Η Μολδαβία το μεταφέρει τώρα το τρίτο ενεργειακό πακέτο θα εγκριθεί πιστεύω από το Κοινοβούλιο μέσα σε ένα-δυο μήνες. Εδώ βρισκόμαστε το μεγαλύτερο πρόβλημα στο μέλλον. Δεν είναι μεταφορά και η δευτερογενής νομοθεσία, αλλά η κωδική δικτύων είναι πολύ σημαντική για την πλήρη εφαρμογή, θα πρέπει να προταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά προβλέπεται και το ζήτημα είναι πώς να συγχωνεύσουμε αυτούς τους ε, κωδικούς από την άλλη πλευρά των συνόρων. Δηλαδή, πώς ε, τα κράτη-μέλη θα συνδράμουν στο συμβατικό πλαίσιο στους εμπλεκόμενους φορείς. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ε, μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη συμμόρφωση. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε δυνάμει του άρθρου 15, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε όλες τις νομικές πράξεις προβλέπεται κάτι τέτοιο. Υπήρχε ένα άλλο ερώτημα για το North Stream 2. Για να απαντήσω αμέσως, γιατί να μας απασχολεί αν υπάρχει πληθώρα φυσικού αερίου. Ίσως αυτό το ε, σχέδιο, το πρόγραμμα να μην ε, είναι ε, αξιόπιστο και να μην είναι βιώσιμο περισσότερο. Νομίζω ότι αυτά τα μεγάλα σχέδια υποδομών έχουν συγχωνευτεί με πολιτικές συνιστώσεις και δυστυχώς ε, δεν είναι οικονομικά βιώσιμα. Αλλά ποιος ξέρει τι θα συμβεί με όλα αυτά τα νομικά ζητήματα. Ίσως η Σενιέρ θα μπορούσε να εξάγει τόσο πολύ ενέργεια στην Ευρώπη έτσι ώστε το Nord Stream 2 να οδηγήσει την Gazprom στην πτώχευση και να ισχύσει κάτι τέτοιο όπως και στην περίπτωση του South Stream. Ας το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ντιφούρ, με τη σειρά θα δω τις ε, ερωτήσεις, θα τις ομαδοποιήσω κάπως. Το κύριο Τόμας... Ε, σε σχέση με τη ζήτηση φυσικού αερίου. Θεωρώ ότι υπάρχει ζήτηση φυσικού αερίου. Το 75% της ζήτησης αφορά έξι χώρες. Θεωρούμε ότι θα υπάρχει μία πτωτική τάση. Δεν αφορά την οικονομική κρίση αφορά τις διαφορετικές αλλαγές στην οικονομία. Η βασική διαφορά με τον ε, διπλανό μου έγκυται στο πόσο φυσικό αέριο χρειαζόμαστε, όχι, όχι πόσο υπάρχει και πόσο έρχεται εκτός Ευρώπης. Το ζήτημα είναι πόσο, πόσες ανάγκες πραγματικών εισαγωγών έχουμε. Υπάρχουν προβολές που δείχνουν αύξηση της ζήτησης στην Ευρώπη. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με σενάρια τα οποία δεν συμβαδίζουν με τα, τις ενεργειακές ανάγκες και τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πόσο φυσικό αέριο χρειαζόμαστε στην τομέα μεταφορών ή πόσο ε, βιοφυσικό αέριο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει πραγματική ανθεκτικότητα, γιατί νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε πολλά στο τομέα των ε, υποδομών. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε επιπρόσθετη ε, προμήθεια, αλλά είναι χαμηλή η αριθμή, δηλαδή λιγότερο από ένα δις. Εάν το συγκρίνουμε με τις αποδομές που προγραμματίζονται μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πληθώρα, αλλά θα έχουμε να κάνουμε με ένα 58% πάνω από αυτό που έχουμε και δεν χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ε, χρειάζεται να δαπανίσουμε τόσο υψηλό κεφάλαιο. Δεν λέω ποιο σχέδιο χρειαζόμαστε και ποιο όχι. Αν δούμε το «North Stream 2, αναρωτιόμαστε πολιτικά κατά πόσο δεν είναι επιζήμιο για την Ευρώπη. Δεν οδηγεί σε διαφοροποίηση χρήσεων και χρήσης και δεν υπάρχει εξορθολογισμός ως προς τη χρήση. Ως προς τη ε, ρήξη παροχής σε συγκεκριμένα δίκτυα και ιδιαίτερα σε σχέση με αυτά που προαναφέρθηκαν, Νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η, μήτος, η μείωση της ζήτησης και αυτό που έχει σημασία είναι αν πραγματικά χρειαζόμαστε περισσότερες ροές. Έτσι ώστε να μην υπάρχει ρήξη και ιδιαίτερα σε σχέση με τα ε, πυρηνικά, σε σχέση ε, με το software και το hardware, αυτό που μας ενδιαφέρει σε σχέση και με τον OPEC είναι να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες. Δεν χρειαζόμαστε νέους ε, αεραγωγούς, αλλά καλύτερη ρύθμιση, κανονιστική ρύθμιση, έτσι ώστε να έχουμε μείωση της ε, ζήτησης, μια ήπια προσέγγιση και όχι τη δημιουργία νέων τερματικών σταθμών. Ο κύριος Άντρου Βόκερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ενδιαφέρουσα η επιλογή των ερωτήσεων. Φυσικά θα είναι θέμα πολιτικής επιλογής στο μείγμα φυσικού αερίου. Εμείς ε, ως ε, εταιρεία φυσικού αερίου θα λέγαμε ότι έχει σημασία να υπάρχει φυσικό αέριο στο μείγμα ως ε, αντιστάθμισμα σε ενδεχόμενο πρόβλημα σχέση με τις ανανεώσιμες έχει χαμηλότερη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, γενικά χαμηλότερες εκπομπές. Πρέπει να έχει λοιπόν μεγαλύτερη συμμετοχή στο μείγμα. Ε, το ότι δεν ε, σχολίασα για το κλίμα ε, οφείλεται στο ότι δεν είχα αρκετό χρόνο στο περιορισμό σε 8 λεπτά της ομιλίας μου. Δεν ήθελα να υπενηχθώ ή αδίποτε αντιπαράθεση μεταξύ των υποστήρικτων του κλίματο και εκείνων που θέλουν να προωθήσουν το φυσικό αέριο και κυρίω το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Απλώ δεν είχα το χρόνο και περίμενα με τι ερωτήσει να δώσω απαντήσει. Εμεί αναπτύσσουμε υποδομέ στι ΗΠΑ. Το μείγμα θα το αποφασίσει βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε παρά να κάνουμε μόνο προτάσει και τίποτα περισσότερο. Είμαστε υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, σε μια παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου. Αυτό θα είναι στόχος πιστεύω της Αμερικανικής κυβέρνησης. υποστηρίζουμε τις προτάσεις ε, της νομοθετικής επιτροπής σας και άλλων, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρεθεί σε θέση να αξιοποιεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό αυτές τις δυνατότητες προσφέρει διαρκώς εξελισσόμενη αγορά φυσικού αερίου, ανταγωνιστικότητα ενισχυμένη στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ασφαλώς θα οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές, είτε πρόκειται για περίοδο ε, ισχνών αγελάδων, είτε πρόκειται για μια ε, προοπτική και ένα σχεδιασμό. Πιστεύουμε ότι ο περιορισμός του ανταγωνισμού, περιορίζοντας και την πρόσβαση ε, και με τον περιορισμό ταυτόχρονα της πρόσβασης σε διεθνείς αγορές φυσικού αερίου, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Και χώρες όπως η Πολωνία, η Λουθωνία και άλλες που έχουν πολύ περιορισμένη ποικιλία προμήθειας φυσικού αερίου βρέθηκαν ε, σε πολύ δινή θέση όταν έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουν ε, προβλήματα στις προμήθειες. Πιστεύουμε λοιπόν, όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε, μια, ε, σε ένα καλύτερο μείγμα. Σε σχέση με τις τιμές και τη συγκεκριμένη ερώτηση που διατοπίθηκε, δεν θα επισέλθω στις συγκεκριμένε ερωτήσεις σας, αλλά θα σας δώσω μια γενική εικόνα που υποστηρίζει πιστεύω τα όσα είπα. Οι εξελίξει σχέση με την προμήθεια, οι χαμηλέ τιμέ των βασικών προϊόντων στην αντικυκλική αυτή περίοδο έχουν οδηγήσει και σε χαμηλέ τιμέ φυσικού αερίου οι υποδομέ φυσικού αερίου που έχουν αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό του, τα πρόκειται για αγωγού, τα πρόκειται για τερματικά υγροποιημένου ε, αερίου, βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο κόστου. Μπορούμε ταυτόχρονα όμω να προσφέρουμε φυσικό αέριο πολύ πρόθεσμα και σε πολύ χαμηλέ τιμέ, με 4,50 4,5 δολάρια. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι το αγωνιστικό σχέση με τι υφιστάμενε τιμές. Είδαμε άλλωστε πρόσφατα άφηξη τέτοιων φορτίων στην ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα, εάν υπάρξουν επιπλέον υποδομές προμήθειας αερίου, θα πρέπει να κοιτάξουμε μακροπρόθεσμα. περιθωριακά χαρακτηριστικά της αγοράς και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η ζήτηση για το αέριο στα 7 με 8 δολάρια MBTU. Αυτό που κάνει η, Ευρωπαϊκή, η Αμερικανική προμηθευτική πλευρά είναι η διαφάνεια ως προς τις τιμές και το ότι δηλώνει πως εάν θέλετε αέριο για το μέλλον μπορούμε να δεσμευτούμε σε αυτές τις τιμές και αν ο προμηθευτής σας, ο τακτικός σας ζητήσει υψηλότερη τιμή, τότε στραφείτε, απευθυνθείτε σε εμά και εμείς θα σας εξασφαλίσουμε αυτές τις χαμηλότερες τιμές. Είναι πολύ ισχυρό νομίζω διαπραγματευτικό εργαλείο αυτό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν γνωρίζει ότι μπορεί, ο εναλλακτικό προμηθευτή είτε είναι Ρώσο, νορβηγό, Εγχώριο κτλ. να ε, προσπαθήσει να αυξήσει τις τιμές. Αυτά για τις ε, απαντήσει, αν και δεν είμαι σίγουρη ότι έχω καλύψει όλε τι ερωτήσει, Πρόεδρε. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ. Μα τελειώνει ο χρόνο Δύο ακόμα οι συναδελφοί μου ζητούν τον λόγο για ερωτήσει. Σα παρακαλώ να περιοριστείτε στα 30 δευτερόλεπτα, κύριε Τουρμέση. Όχι, 10 δευτερόλεπτα, Πρόεδρε. Κύριε Βόκερ, τέσσερα λεπτά επιπλέον σα δόθηκαν και πάλι όμω δεν απαντήσετε σε μια πολύ απλή ερώτηση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ε, εκπομπών ανθρακικού ε, περιεχομένου από την υδρορογμάτωση και κλιματικών ε, επιρροών από το φυσικό αέριο. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Από την υδρορογμάτωση, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικότερη η επίδραση στην ε, κλιματική αλλαγή. Ο κύριο Σαφοζέχ, μια ερώτηση μόνο για τι διαφανεί τιμέ που αναφέρατε. Εάν οι τιμέ σα ενσωματώνουν ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η τιμή θα είναι διαφορετική. Εάν ενσωματώνουν την απόσβεση σε 8-10 χρόνια ή 15, πάλι θα είναι διαφορετική τιμή. Άρα δεν έχει καμία σημασία αυτό που μας λέτε. Και η τιμή δεν πρέπει ακριβώς να έχει σαν νόημα να διευκολύνει την ενεργειακή ε, μεταλλαγή. Για να μπορεί δηλαδή να γίνει αυτή η μεταλλαγή η ενεργειακή δεν πρέπει να είναι οι τιμές κατάλληλες κατάλληλα σχηματισμένος ο κύριος Βόκερ για να απαντήσει. Κοιτάξτε. Τιμολόγηση και άλλες πτυχές των διαφορών καυσίμων. Νομίζω ότι τα πάντα εξαρτάται από την πολιτική της αγοράς. Πώς θέλει δηλαδή να ορίσει και να προχωρήσει. και πλεονεκτήματα υπάρχουν και μειονεκτήματα σε κάθε περίπτωση. Και οι φόροι που θα επιβληθούν μπορεί να ευνοήσουν μια επιλογή έναν τον άλλον. Εμείς είμαστε ε, επιχείρηση ανάπτυξη υποδομών στις ΗΠΑ. Δεν νομοθετούμε. Ε, δεν υποδεικνύουμε φόρους στην προϊόντα για το σχιστολιθικό αέριο. Αναπτύσσουμε, όπως είπα, υποδομές εμείς δεν παράγουμε φυσικό αέριο στο ισχυστολιθικό αέριο στις ΗΠΑ. Αλλά θα μπορούσα να υποδείξω κάποιες ε, έρευνες που αναφέρονται σε χαμηλότερες εκπομπές, πέραν των οποίων όμως δεν μπορώ να δώσω όλες λεπτομέρειες. Πάντως, στις ΗΠΑ η παραγωγή γίνεται με βάση την κρατική ή ομοσπονδιακή ε, νομοθεσία για την υδρορογμάτωση ώστε να παράγεται αυτό το συστολιθικό φυσικό αέριο όπως το ε, επιθυμεί, όπως το ορίζει η κυβέρνηση κάθε φορά. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να προσθέσω. Καλώς λέω πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτή τη μία ώρα και κάτι. Τώρα πάμε στο δεύτερο μέρος που αφορά την Ενεργειακή Ένωση και την ελεύθερη αγορά. Φίλοι εχθροί, θα ήθελα Θα ήθελα και οι δύο μιλητές να αρκεστούν στα 8 λεπτά. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Ντεσκάλτσι. Ο κύριος Κλάουντο ε, Δεσκάλση, ο οποίος ήταν ε, εκτελεστικός διευθυντής της ΕΝΗ. Ή και είναι, ήταν και είναι. And, uh, well, you joined ENI uh, ε, some years ago. Και από όσο γνωρίζω, Ενταχθήκατε στην ε, ΕΝΗ το 1981, είχατε πολλές διευθυντικές ε, θέσεις και ήσασταν και εκτελεστικός αντιπρόεδρος για διάφορες περιοχές ε, ανά τον κόσμο. και ήσασταν πρόεδρος της ΕΝΗ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο πρώτος Ευρωπαίος ε, στον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου που ε, λάβατε ένα τιμητικό μετάλλιο, ε, το μετάλλιο Charles Rand το 2012 και είσαστε και μέλος του Δικητικού Συμβουλίου της Κομφιντούστρια. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε τη δική σας ε, εισήγηση. Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Μπούζεκ για αυτή την ε, ε, ευγένεια του, για την ευγενή του πρόσκληση και θα ήθελα να συζητήσουμε για θέματα που άπτονται της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό είναι ένα ζήτημα ζωτικής ε, σημασίας για την Ευρώπη που είναι καθαρός εισαγωγέας. Το 2000 ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρήγε πάνω από 50% των αναγκών σε φυσικό αέριο. Τώρα έχει μια πτωτική τάση, δηλαδή έχει φτάσει στο 30% και σε λίγα χρόνια θα βρισκόμαστε κάτω από το 20%. Γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη ε, ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ενέργειας. Επίσης είναι επίγουσα σημασίας η δημιουργία ενός βιώσιμου και διαφοροποιημένου ενεργειακού μείγματος και επίσης να υπάρξει και μόχλευση των τεράστιων επενδύσεων που έχουν γίνει μέχρι τούδε. Από τη δεκαετία του 70 η Ευρώπη στρατηγικά επέλεξε να βασιστεί στο φυσικό αέριο ως τον πιο καθαρό και αξιόπιστο καθώς και αποδοτικό ε, ενεργειακό μείγμα και πηγή. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο κρίναμε ότι θα πρέπει να βασιστούμε στους ε, διάφορους, ε, στις διάφορους οδούς παροχής ενέργειας. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία γιατί με τη χρήση φυσικού αερίου μπορούμε να μειώσουμε στο μισό τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με τη χρήση του άνθρακα. Τώρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές υποδομές στον κόσμο με τη δυνατότητα εισαγωγής ενός 60% σε σχέση με την τρέχουσα ζήτηση, δηλαδή 465 BCM παραγωγικής ικανότητας παροχής μέσω αγωγών και 200 ε, BCM σε σχέση με παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Έτσι, ε, τα τελευταία 20 χρόνια μπορέσαμε να επενδύσουμε πάνω από 65 ε, δις ευρώ σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα στον τομέα του φυσικού αερίου με βάση ε, μία εισαγωγική ικανότητα της τάξης του 40% και αποθήκευσης 50%. Επίσης, μπορέσαμε να έχουμε ε, να οικοδομήσουμε νέες μονάδες που μπορούν να καλύψουν ανάγκες 150 GB gigabyte και να gigawatt με συγχωρείτε και να φτάσουμε σε μία δαπάνη της, της τάξης των 240 δις. Αυτό αφορά και την αύξηση της ζήτησης κατά 30% στην περίοδο μεταξύ 2000 και 2009. Όμως δυστυχώς μετά υπήρξε μία πτωτική τάση και μειώθηκε η ζήτηση στα 400 BCM το 2014 και μειώθηκε ο κύκλος, ο συντονισμένος κύκλος ε, υποδομών σε 45% και στη συνέχεια σε 30%. Από το 2008 και μετά η Ευρώπη ήταν η μοναδική ήπειρος που μπόρεσε να ορίσει στόχους πρόκληση με βάση την επιδότηση, τη μεγάλη επιδότηση και των ανανεώσιμων. Το 2014 οι επιδοτήσεις ανήλθαν σε 75 δις δολάρια που αντιστοιχεί στο 55% των παγκοσμίων επιδοτήσεων στις ανανεώσιμες. Αυτό αφορά και το ενεργειακό μείγμα, κάτι το οποίο αποτελεί μια, ένα πραγματικό παράδοξο. Δηλαδή, το, τα τελευταία χρόνια οι ανανεώσιμες έχουν αναπτυχθεί κατά 8%. Όμως αυτή η ανάπτυξη ακολουθήθηκε και από τη χρήση άνθρακα, κάτι το οποίο αποτελεί ένα πραγματικό παράδοξο. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε σε μια σωστή επιδότηση των ανανεώσιμων, ε, μιλώντας για ένα μερίδιο 25% στην Ευρώπη μέσα στα πλαίσια του ενεργειακού μείγματος, δημιουργώντας ένα 76% εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι μειώσαμε και τα ευεργετήματα που απορρέουν από τις ανανεώσιμες. Δηλαδή, στην ουσία εξουδετερώνουμε τα ευεργετήματα από τη χρήση του 10% των ανανεώσιμων. Επίσης, ο άνθρακας ήταν η μόνη λύση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες προμήθειας. Ως προς το πρώτο θέμα, ο περιβαλλοντικός στόχος έχει ένα ενεχόμενο κόστος και αυτό έχει επιπτώσεις και στον πλανήτη και στη ζωή μας. Ως προς το ενεργειακό μείγμα όμως θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή στο δεύτερο θέμα, δηλαδή την ασφάλεια και διαφοροποίηση προμήθειας φυσικού αερίου. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις, ε, στη μελλοντική ζήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, πέρα από τους ε, παραδοσιακούς προμηθευτές, δηλαδή τη Νορβηγία, τη Ρωσία και την ε, Αλγερία, θα μπορέσουμε να έχουμε νέους ε, γίγαντες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ανατολικής Αφρικής. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι το δέλτα του Νείλου θα μπορέσει να ε, χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει αυτό το δυναμικό σε σχέση με τις πηγές που έχουν ανακαλυφθεί στη Λιβύη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα ακολουθήσει μία νέα οδό προς την Ευρώπη με μείωση των τιμών. Αυτό αφορά και την προμήθεια από τις ΗΠΑ. Γι' αυτό ακριβώς η ε, προμήθεια φυσικού αερίου είναι πιο ασφαλής, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική σε σχέση με το παρελθόν. Ε, δεν μπορούμε να αφιστούμε μέσον έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το πρότυπο ενεργειακής ασφάλειας μέσα στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης αγοράς φυσικού αερίου, εάν λάβουμε υπόψη και τους στόχους για το 2030 που όρισε η COP21. Οι ανανεώσιμες ε, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και συνοδευτικά μέτρα και μέσα, έτσι ώστε να έχουμε μία ε, συνεχή βιώσιμη λύση. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε στο φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες έτσι ώστε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα και να έχουμε μία αγορά η οποία να ε, παρέχει, να προβάλλει αυτή την προμήθεια η οποία θα είναι αξιόπιστη, ανταγωνιστική και διαφοροποιημένη. Έχουμε αναγνωρίσει τους ε, διάφορους τομείς και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι από το 2000 και μετά θα πρέπει να προωθήσουμε την παραγωγή της εγχώριας αγοράς. Ορισμένες χώρες μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή και αυτό θα ε, οδηγούσε στη μείωση της εξάρτησης από τις ε, εισαγωγές. Και το δεύτερο σκέλος αφορά την διασυνδεσιμότητα Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί στη μεταφορά φυσικού αερίου από την ε, Ισπανία στη Γαλλία, από την Ιταλία στη Γερμανία και από τη Γερμανία στις ε, ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει όμως να υπάρχει διασυνδεσιμότητα υποδομών έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μεγάλο δυναμικό στα δύο κομβικά σημεία της Ιταλίας και της Ισπανίας. Έτσι θα μπορέσουμε να ε, ανταποκριθούμε στα πλαίσια κερδών και μέσα στα πλαίσια του ρυθμιστικού πλαισίου θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα διεθνικό εμπόριο για να ανταποκριθούμε και στην τιμολόγηση. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Θα πρέπει όμως να έχουμε μια ενιαία αγορά έτσι ώστε να κινηθούμε και πέραν αυτής να οικοδομήσουμε ένα ενεργειακό μοντέλο το οποίο να βασιστεί στο φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες με βάση τις παραγωγικές ικανότητες της τελευταίας δεκαετίας. Έτσι θα μπορέσουμε πραγματικά και αποδοτικά να μειώσουμε τις εκπομπές με βάση μια βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη για την Ευρώπη. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κλάουδιος Κάλτσι πρέπει να φύγει σε 5-10 λεπτά. Γι' αυτό ε, ε, θα ήθελα να ε, πάρω κάποιες σύντομες ερωτήσεις. Πρώτος έχει καταγραφεί ο κύριος Μενσεν. Thank uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση σε σχέση με την αγορά αερίου στην Ευρώπη. Συζητήθηκε και από το πρώτο πάνελ το θέμα του Nord Stream 2. Ξέρουμε ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε την προμήθεια αερίου στην Ευρώπη. Αλλά πώς να σας το πω. Μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια, για ασφάλεια προμήθειας. Αλλά ακούμε και από το πάνελ ότι θα χρειαστούμε πολλά κυβικά μέτρα στο μέλλον. Και για την ώρα δεν έχουμε ενεργειακή ένωση και οι χώρες μπορούν να πάρουν ξεχωριστές αποφάσεις καθεμία για τον εαυτό της. Ας πούμε η Γερμανία και η Ρωσία μπορούν να αποφασίσουν από μόνες τους ε, για το πώς ε, θα αγοράσουν. Ε, έχουμε το EDA που κάνει τα δικά του. Επομένως, ποια είναι η άποψή σας, αυτό ρωτώ, ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με το ε, τι μπορούμε να κάνουμε για το Nord Stream 2. Δηλαδή θέλετε να με ρωτήσετε ποια είναι η άποψή μου για το Nord Stream 2. Ωραία. Ο κύριος Τζανονάτο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ε, τον εκτελεστικό διευθυντή της ε, ΕΝΗ που δέχτηκε σήμερα να έρθει εδώ να συναντηθεί με την Επιτροπή μας. Ε, συμφωνώ σχεδόν με όλα αυτά που μας είπε. Η σημασία του ε, φυσικού αερίου, του μεθανίου, ε, η ανάγκη διαφοροποίησης των υποδομών, όλα αυτά τα συμμερίζομαι. Ερώτηση. Το παρόν κόστος του, του πετρελαίου, με ποιο τρόπο έχει επίπτωση στην αγορά φυσικού αερίου. Ένας από τους ε, λόγους που συχνά αναφέρεται ε, για τις ε, περιπτώσεις αυτές είναι η προσπάθεια από τις αραβικές χώρες, Σαουδική Αραβία κλπ. να πολεμήσουν την, το, το αέριο, να, να μην το αφήσουν να φτάσει στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τούρμες. Εγώ σας ευχαριστώ είπατε ότι οι ανανεώσιμες πηγές δημιουργούν προβλήματα. Ε, μιλάτε, αναφέρεστε στο, στις επιδοτήσεις, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα των, της μόλυνσης ε, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των ε, επιδοτήσεων. τώρα βλέπουμε συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες δεν αφορούν το κλίμα ε, αλλά αφορούν ε, εσωτερικές αποφάσεις σε σχέση με το πετρέλαιο. Είχα μία την χαρά μαζί με την κυρία Μποναφέ να ε, προεδρεύσω σε μία συνεδρίαση ε, που ασχοληθήκαμε ακριβώς με ε, αυτά τα ε, ζητήματα. Μήπως εσείς μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια περισσότερα όσον αφορά την στρατηγική. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντεσκάλτσι. Αναφερθήκατε σε πολλά και σημαντικά θέματα για την Συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο κύριος Δεσκάλτση, δεν γνωρίζω τη γλώσσα σας, θα πρέπει να βάλω Ε, να βάλω λοιπόν τα ακουστικά μου. Αναφερθήκατε σε δύο σημαντικά θέματα όσον αφορά ε, την ε, ασφάλεια της προμήθειας από τη μία ε, του, του αερίου, από τη μία την εσωτερική παραγωγή η οποία θα πρέπει να προωθηθεί βάση της, ε, ε, των διασυνδέσεων, αλλά αναφερθήκατε και σε ένα νέο φαινόμενο, κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, ε, που αφορά επίσης την εσωτερική παραγωγή, που θα μπορούσε δηλαδή να έχει επίπτωση στην εσωτερική αγορά, αναφέρομαι στην Κύπρο αλλά στα πλαίσια μικρότερης ε, τιμής, χαμηλότερης τιμής ε, του αερίου, ποια είναι η εκτίμηση που κάνετε ε, σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, πώς μπορεί να προωθηθεί δηλαδή το φυσικό αέριο που θα παραχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, όσον αφορά τις υποδομές, την ενδυνάμωση των διασυνδέσεων κτλ. Όλα αυτά είναι προγράμματα ε, ε, πολύ σημαντικά. Ε, συμφωνείτε με αυτό. Η υποδομή στην Νότια Ιταλία, ας πούμε, είναι αρκετή. Οι μηχανισμοί διασύνδεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλές. Η κυρία Τόια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Εσείς αναφερθήκατε κυρίως στο θέμα της ε, ε, ασφάλειας αλλά και της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας που είναι δύο κύριοι στόχοι της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ιδιαίτερως αναφερθήκατε σε ένα σημείο το οποίο επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, η, ε, λόγω των ε, λοιπόν πόρων για μεγαλύτερες επενδύσεις εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει. Οι διασυνδέσεις κατά την άποψή σας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερο γιατί είναι ακριβώς περιουσιακά στοιχεία τα οποία ήδη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γιατί κινδυνεύουμε να έχουμε μια διπλή, ένα διπλό παράδοξο, δηλαδή και λιγότερα, λιγότερους πόρους, αλλά και ε, λιγότερη χρήση των ε, διασυνδέσεων και των υποδομών. Η κυρία Μποναφέ, ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεσκάλτσι. Δεν θέλω εγώ να υποβιβάσω την σημασία του αερίου όσον αφορά την επίτευξη στόχων βάσει της τελευταίας κόπ του Παρισιού ή να υποτιμήσω την αξία όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Ε, εσείς αναφερθήκατε σε διάφορα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν κύρια στοιχεία της ενεργειακής πολιτικής, δηλαδή διαφοροποίηση των πηγών και διαφοροποίηση των διαδρομών. Εμείς έχουμε συζητήσει πολλές φορές τα θέματα αυτά και ε, πολλοί ε, ευρωβουλευτές ε, έχουν αναφερθεί και στο θέμα του Nord Stream 2, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και το δυναμικό της Μεσογείου, θα ήθελα την άποψή σας σχετικά με τη δημιουργία ενός κόμβου, ενός hub στην Μεσόγειο, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η εισαγωγή αερίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Στρέφομαι σε εσά κύριε Ντεσκάιτσι ε, και σας ζητώ να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε. Οι τιμές του αερίου και το Nord Stream 2. Όπως ξέρετε δεν είμαστε στο Nord Stream 2 ο Nord Stream 2 είναι ε, αγωγός για τη Βόρεια Ευρώπη. Στην Ολλανδία υπάρχει μείωση της παραγωγής αερίου, άρα χρειάζονται, οι, οι ανάγκες είναι αυξημένε. Η επίπτωση του Nord Stream 2 σημαίνει ότι θα βάλουμε περισσότερο αέριο εκεί, άρα θα δημιουργήσουμε ένα ισχυρότερο κόμβο στο βορρά και θα δημιουργήσουμε ε, επομένως υψηλότερη τιμή για την νότια ας πούμε Ιταλία εάν το αέριο δεν έρχεται απευθείας από την ε, Ρωσία γιατί η τιμή μεταφοράς θα αυξηθεί, το κόστος μάλλον μεταφοράς θα αυξηθεί μεταφοράς προς την Νότια Ευρώπη. Άλλη ερώτηση. Πετρέλαιο έναντι αερίου. Νομίζω ότι οι τιμές του αερίου ακόμα σχετίζονται, διασυνδέονται με το πετρέλαιο, όχι παντού. Ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, ε, δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση ανάμεσα στις τιμές ε, αερίου και πετρελαίου. Στην Ευρώπη, όμως, ήδη ε, συγγνώμη, εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει η διασύνδεση. Έχουμε αέριο από τη Ρωσία, από την Νορβηγία, από την ε, Αλγερία. Εξακολουθεί να υπάρχει τέτοια διασύνδεση. Κόμβος ε, αερίου στην η αυξάνονται και στο βορρά και στο νότο και εκεί δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση με τις τιμές ε, του ε, πετρελαίου. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε ε, τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια και με τη Ρωσία και με την Ορβηγία. γιατί είδαμε ότι όταν το πετρέλαιο ήταν ε, ε, ψηλά, ε, το αέριο ήταν πιο χαμηλά. Εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρώπη διασύνδεση ανάμεσα στα δύο αυτά καύσιμα. Στον ειρηνικό υπάρχει ακόμα διασύνδεση και μάλιστα 100% υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στο αέριο και το πετρέλαιο. Όσον αφορά τώρα την άλλη, την επόμενη ερώτηση. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως. Είπα σαφώ ότι ό,τι ξοδεύουμε σε ε, ανανεώσιμες ε, πρέπει να τα ξοδέψουμε. Καλά κάνουμε. Δεν είπα ότι δεν είναι μακροπρόθεσμη αξία για τον πλανήτη ή για τον άνθρωπο. Δεν τίθεται να αμφιβόλω αυτό. Αυτό το επιχείρημά μου όμως είναι διτό. Πρώτον, ότι τις τελευταίες δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεσε προς το ε, αέριο και επομένως οι βιομηχανίες ε, έκαναν τεράστιες επενδύσεις κατά την έφθηση αυτή ε, και δημιουργήσαμε εν τέλει ένα παράδοξο γιατί από τη μία πλευρά επενδύσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια 200 δις ευρώ για να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες και πολύ καλά κάναμε γιατί αυτό στρέφεται προς το μέλλον, αλλά ταυτόχρονα και από την άλλη πλευρά δεν προσέξαμε το ενεργειακό μείγμα. Και εν τέλει, εάν ε, ε, βάλει κανείς χρήματα και προσπάθειες μακροπρόθεσμα στις ανανεώσιμες πηγές ε, είναι καλό, αλλά εάν ταυτόχρονα δεν ελέγχει κανείς και το ενεργειακό μείγμα προκύπτει ισχυρό παράδοξο και αναφέρομαι στην ενέργεια γενικότερα και όχι μονάχα ε, στην ηλεκτρική ενέργεια. Ε, η χρήση του άνθρακα αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια ε, γιατί το κόστος της ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό στην Ευρώπη. Γιατί το ε, κόστος της ε, ενέργειας ε, είναι στην ουσία τριπλάσιο από το κόστος της ενέργειας το αντίστοιχο στην, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και επομένως ε, ε, λόγω ακριβώς της χαμηλής τιμής ε, που είχε το, ο άνθρακας στα τελευταία χρόνια, αυτό οδήγησε σε μια τάση αποθήκευσης και αγοράς άνθρακα με αποτέλεσμα να αυξηθεί εν τέλει η χρήση του και να βαρύνει περισσότερο στο ενεργειακό μείγμα. Ε, αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο ε, για το ενεργειακό μείγμα ε, και μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα ε, είναι να ε, υπάρχουν, να εφαρμοστούν περιορισμοί όσον αφορά τις εκπομπές και όσον αφορά ε, τις χρήσεις στα διάφορα εργοστάσια. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, ας πούμε, έχουμε συγκεκριμένη επιδότηση όσον αφορά την παραγωγή εκεί θα πρέπει να μπουν όρια. Και μόνο τότε θα δούμε ότι και το κοκ και ο λιγνίτης και ο, ο άνθρακας και το πετρέλαιο θα χρησιμοποιηθούν λιγότερο. Βλέπουμε ότι κάποιες τράπεζες τώρα δίνουν ε, και ε, δάνεια χρησιμοποιώντας ε, τα εργαλεία EPS. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και από τη μία μεριά να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε πιο αποτελεσματικά εργοστάσια ενέργειας παραγωγής ενέργειας όσον αφορά τον Ανατολικό Κόμβο East Hub είπα, επενδύσαμε πολύ στις υποδομές. Η Ευρώπη δεν έχει πολλούς πόρους. Δεν έχουμε, πολύ... δεν έχουμε αέριο, έχουμε βέβαια ε, αέρα, αεολική ενέργεια. Τέλος πάντων, ε, υπάρχει ζήτημα όσον αφορά ε, την ε, ενεργειακή ασφάλεια, αλλά έχουμε και μία δύναμη. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε, δίνουμε πολλά χρήματα για τις ε, υποδομές. Αυτό, αυτή είναι η δύναμή μας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αέριο, το οποίο παράγεται κοντά στα σύνορά μας. Ο κόμβος Ανατολικής Μεσογείου, ας πούμε. Έχουμε στην Κύπρο, ε, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ 300 BCM ε, αερίου με δυνατότητα διπλασιασμού. Άρα εδώ δημιουργούνται hubs τα οποία όχι μόνο συμπληρώνουν το ένα το άλλο, αλλά ε, και ε, μεγαλώνουν, την, αυξάνουν την ασφάλεια της Ευρώπης. Γιατί μπορούμε πλέον να έχουμε αέριο το οποίο να μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη με ένα λογικό κόστος μεταφοράς. Και εδώ προκύπτει και το ζήτημα των διασυνδέσεων. Οι διασυνδέσεις ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ε, οι υποδομές στην Ιταλία, στην Ισπανία ε, πρέπει να είναι σε θέση να είναι τόσο δυνατέ ώστε να μπορούν να παραδώσουν αέριο στον βορρά. Να αλλάξει δηλαδή πλέον η ροή και να είναι από τον νότο προς τον βορρά. Η αντίστροφη ροή ε, από την Ιταλία προς τη Γερμανία, προς την Αυστρία ε, ε, πρέπει να βελτιωθεί κατά 20 BCM. Αυτό έχει γίνει στην Ιταλία. Είμαστε λίγο ακόμα πίσω στην Ισπανία. Μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας πάντως και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές Βρισκόμαστε κάπου μεταξύ 70 και 90 BCM που μπορούμε να παραδώσουμε στο βορρά. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και το, ε, την εκκίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Είχαμε μέχρι τώρα διαδρόμους ε, ε, κατακόρυφους από βορρά προς νότο. Τώρα πρέπει να δημιουργηθούν και ε, ε, άλλοι διάδρομοι από δυτικά προς τα ανατολικά. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και υποδομές οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε επίση ένα καλύτερο μείγμα. Γιατί τώρα έχουμε περισσότερου πόρου, Είμαστε σε πολύ καλή θέση έχουμε το αέριο το οποίο ε, παράγεται κοντά μας, Βόρεια Αφρική, Μεσόγειο ε, και νομίζω ότι αυτό είναι ε, καλό για το μέλλον και μπορεί να αποτελέσει μια ικανοποιητική λύση για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε μάλλον, Κλάουδιο Δεσκάλτση. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ για να απαντήσετε και τις ερωτήσεις. Δεν σας πρόφερα καλά, λέγομαι Δεσκάλτση, λέει ο μιλητής. Σας ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ. και πάλι. Και τώρα πάμε στον επόμενο. Στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Γκάτα του Στραχώτα. Ασφάλεια, προμήθεια σε αέριο, διαφορετική κίνδυνη, συμφέροντα, εργαλεία προτείνονται. Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωση. 50 χρόνια λοιπόν έρευνα ε, στην αγορά του αερίου, 15 χρόνια εμπειρία στην αγορά αερίου, κυρίως ε, Κασπία, Τουρκία, Ιράν, ε, ενεργειακό Γραφείο Ενεργειακής Πολιτικής της, του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών, όσο υπήρχε, Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχέσεις ενεργειακές, σχέσεις με το φυσικό αέριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας Ουκρανίας, Think Tanks, σχέδια και έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικές πτυχές στην ενεργεια των οριακών τομέων, παραδείγματι, και έχετε συμμετάσχει και έχετε οργανώσει διάφορες διασκέψεις, σεμινάρια των Ευρωπαϊκών Οργάνων, του ΝΑΤΟ, της Διεθνούς Ενεργειακής Υπηρεσίας των Παρισίων και σας παρακαλώ να μας δώσετε το λόγο σας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνετε να σα μιλήσω εδώ για την ασφάλεια στην προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα την ε, διαφοροποίηση και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ε, υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα της προμήθειας σε φυσικό αέριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που αφορούν ε, την προμήθεια σε αέριο της Ένωσης του, οι κίνδυνοι ε, σε σχέση με διατάραξη των ε, προμηθειών σε αέριο από την Ρωσία που ιδιαίτερα ε, κινητοποίησαν να αντιδράσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και άλλα προβλήματα, είτε μετατοπίσεις διαδρομών, είτε διαταραχές στη Βόρεια Αφρική, Λιβύη, Αλγερία, επιτάχυνση της μείωσης της παραγωγής κατά χώρες Δανία και βέβαια πρόκληση είναι και η πιθανή μη βιωσικομότητα των επιπέδων παραγωγής φυσικού αερίου της Νορβηγίας. Ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το τι θεωρούν ε, κύριο κίνδυνο προτεραιότητας και τι μπορούν ή τι θέλουν να πράξουν για να ε, προστατευτούν εναντί πιθανών κινδύνων. Για να δείξουμε λοιπόν αυτές τις διαφορές θα σας παρουσιάσω μια προσεκτική ίσως ε, σύγκριση στάσεις εναντί της ασφάλειας σε προμήθεια αερίου μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας. Στη Γερμανία λοιπόν μακροπρόθεσμα βλέπουμε να εστιάζεται στις, ε, στην αηφορία, στη βιωσιμότητα των εισαγωγών της αλλά και βραχυπρόθεσμα να αναζητεί ένα διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Ε, σε σχέση με το ρωσικό αέριο. Η Γερμανία, οι γερμανικές εταιρείες ε, αναζητούν σταθερότητα και ασφάλεια προμήθειας, αναζητούν στο βαθμό του δυνατού την το χαμηλότερο κόστος, θεωρούν ότι είναι χαμηλότερο το κόστος της Ρωσίας προμηθευτή και βλέπουν κάποια συγκεκριμένα οικονομικά ωφέλη σε σχέση με την προμήθεια από τη Ρωσία σε αέριο και βλέπουμε έναν ενισχυμένο ρόλο της Γερμανίας στην ευρωπαϊκή, στον ευρωπαϊκό χάρτη αερίου. Στη σχέση με τη Ρωσία τίνουν προς την ομαλοποίηση, στις προτεραιότητες ε, πολιτικής έκτακτης ανάγκης, SOS δηλαδή, αναζητούν σταθερούς και αναπτυσσόμενους, αυξανόμενους όγκους ρωσικού αερίου ε, και για το ρόλο της ευρωπαϊκής κοινότητας αναζητούν ε, την υλοποίηση των γερμανικών πολιτικών ε, και επιλογών. Τώρα στην Πολωνία βλέπουμε να υπάρχει μια βραχυπρόθεσμη και μέσοπρόθεσμη ε, διακινδύνευση με σαφή κίνδυνο διαταραχής, αβεβαιότητα στο κατά πόσον μπορεί μακροπρόθεσμα να ενισχυθεί το, ο ρόλος του αερίου στο ενεργειακό μείγμα. Ως προς τη Ρωσία θεωρείται ότι είναι πιθανή πηγή αβεβαιότητας. Ε, ιστορικά η μη τι θεωρείται ότι είναι ακριβώς προμηθευτής αερίου εφόσον βρίσκεται σε ε, δεσπόζουσα θέση στην αγορά της Πολωνίας με συνέπειες όχι μόνο στην αγορά του αερίου αλλά και στην πολιτική, την εξωτερική και την πολιτική ασφάλειας. Η Πολωνία λοιπόν είναι πιο επιφυλακτική ως προς το όραμα για τις σχέσεις με τη Ρωσία στο φυσικό αέριο και προσδιορίζει όρους ε, για τη συνέχιση των σχέσεων αυτών, παραδείγματι την κατάσταση στην Ουκρανία, στη διαφοροποίηση ε, για να αντιμετωπίσει τους έκτακτους κινδύνους, κατάσταση SOS, ε, δίνει ιδιαίτερη έμφαση με τρει διαφορετικές πηγές, όπου μειούται το μερίδιο του ρωσικού αερίου στο μείγμα ενέργειας της Πολωνίας και έχει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα βοηθήσει στην διασφάλιση ενό ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις σχέσεις σχετικές με το φυσικό αέριο, με τη Ρωσία και την Gazprom συγκεκριμένα. Βλέπετε λοιπόν μια διαφοροποίηση σχέσεων και θεωρήσεων. Ίσως αυτό έχει να κάνει και με μια διαφορετική κατάσταση μεταξύ Κεντρική Ανατολική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, αλλά και, ε, μεταξύ, και με διαφορέ στα εργαλεία και τι υποδομέ που αναπτύσσονται Νέες λοιπόν ε, υποδομές, νέα εργαλεία με τους νέους αγωγούς, με τον Nord Stream. Κοινά έργα που υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη, οι εταιρείες και η Gazprom που επιδιώκουν μεταξύ άλλων να εξασφαλίσουν ε, ασφαλές, ασφαλείς προμήθειες ενέργειας, φυσικό αέριο στις τοπικές και περιφερειακές αγορές με πρόσθετους ε, διάβλους ε, μεταφοράς αερίου από τη Ρωσία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ε, ο Nord Stream 1 και 2 μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βόρειο-δυτική και Κεντροανατολική Ευρώπη και χρειάζεται λύση περιφερειακού χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα έργο αμφιλεγόμενο που διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει προβλήματα ε, τα οποία θα πρέπει να περιφερειοποιηθούν, λυθούν σε περιφερειακό επίπεδο και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι δεν ε, ε, υποτάσσεται σε επιλογές και προτεραιότητες κάποιων κρατών ή και εταιριών της περιοχής. Υπάρχουν φόβοι δηλαδή ότι μπορεί να ενισχυθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, και να ενισχύσει την θέση της Gazprom στην, στις εθνικές αγορέ. αγορές. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε ε, συνέπειες σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και βέβαια υπάρχει και αβεβαιότητα σε σχέση με την τήρηση του ευρωπαϊκού ε, νομοθετικού πλαισίου. Υπάρχει τώρα η δεύτερη ομάδα έργων που αποσκοπούν στην ασφάλεια μέσω της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας. Ο στόχος συνήθως είναι να ενισχυθεί να μειωθεί η εξάρτηση από τη μία πηγή τη Ρωσία συνήθως και γι' αυτό συνήθως βλέπουμε να υποστηρίζεται από ορισμένα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αυτή η διαφοροποίηση και ταυτόχρονα ε, στοχεύεται και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ενοποίηση τοπικό και περιφερειακό επίπεδο των αγορών Επαραδείγματι, ο νότιος αγωγός φυσικού αερίου, το ε, πρόσφατα ανανεωμένο έργο Βαλτικού, ε, στη Βαλτική από την Νορβηγία, αλλά και για τη Βαλτική και την Αδριατική θάλασσα. Βλέπουμε έργα μικρότερα επίσης ε, σε ε, εύρος, ε, σημαντικά για ορισμένες και μία μόνο χώρες, ε, χωρίς όμως απαραίτητα σημαντικό αντίκτυπο σε περιφερειακό επίπεδο. Δυσκολία στην υλοποίηση είναι τα εμπόδια στην είσοδο στην αγορά με την εγκαθιδρυμένη ε, δεσπόσα θέση της Γκάσπρο, όπως βλέπουμε σε ορισμένες περιπτώσεις, ε, ο σχεδιασμός για την προμήθεια μικρών και κατακαιρματισμένων αγορών και γι' αυτό χρειάζεται υποστήριξη και πολιτική και συντονισμός για να προχωρήσουν τα σχέδια αυτά. Παράλληλα με αυτά λοιπόν έχουμε μια ευρωπαϊκή πρόταση ένα πακέτο μετρών για τον χειμώνα, για το φυσικό αέριο και ανανεωμένος κανονισμός κατά της ανάγκης SOS. Στόχος είναι η αναβάθμιση ενός κοινού ε, συνόλου μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νέες προτάσεις ε, με νέες περιφερειακές ομάδες, ενισχυμένο ρόλο περιφερειακού σχεδιασμού αλληλεγγύης, πλατφόρμες από διάφορες ομάδες ή ομάδες χωρών, ε, Κεντροανατολική Ευρώπη, Βορειοδυτική Ευρώπη, Γερμανία, Πολωνία, που μπορούν έτσι να συνομιλούν μέσα από τις πλατφόρμες και να ορίζουν προτεραιότητες και να εξηγούν τους λόγους ε, της διαφοροποίησής τους. Ενδεχομένως από εκεί θα προκύψουν και οι υποχρεώσεις για την εξέβρεση κοινών περιφερειακών λύσεων με έναν τουλάχιστον κοινό στόχο και ίσως μπορεί αυτό να οδηγήσει και σε μια διάχυση των βέλτιστων πρακτικών στι περιοχές αυτές. Έτσι μπορεί να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά, να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη και να ανοικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με προβλήματα στην προμήθεια. Βέβαια η πρόταση μπορεί να οδηγεί και σε κάποια ερωτηματικά σε σχέση με την ελληνική και την επικουρικότητα, πώ θα ε, επαναπροσδιοριστούν οι τοπικέ περιφερειακέ προτεραιότητες για την αγορά εργασία και την προμήθεια του αερίου, ποια είναι η σχέση μεταξύ της προμήθειας, της ασφάλειας σε προμήθεια και της αγορές, πώς μπορεί αυτή δηλαδή να επηρεάσει σε, περιοχές, σε περιόδους όπου δεν υπάρχει εκτακτή ανάγκη την, ε, τους μηχανισμούς ε, διάθεσης του αερίου και με συγχωρείτε που μακρηγορώ. Ε, έχουμε λοιπόν σαφείς διαφοροποίησεις και αποκλείς μεταξύ κρατών μελών σε διάφορους τομείς, στόχους και εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σαφής η ρόλη των διαφορών παραγόντων, φορέων και θεσμικών οργάνων. Αυτό εμποδίζει το σχεδιασμό κοινή αποτελεσματικής πολιτικής για την ασφάλεια στην προμήθεια του ε, φυσικού αερίου ή για κάθε πολιτική για την ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελευταία ανάλυση και την αποτελεσματικότητα των παραγόντων και φορέων και βέβαια αυτό μπορεί να έχει και συνέπειες προς την εξέλιξη των μέσων που θα ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντιμετώπιση κατά των αναγκών. Ευχαριστώ πολύ και σας συγγνώμη. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σωστακόβα γιατί μας κάνατε μία πολύ σωστή κυρία Στραχώτα. Μας κάνατε μία πάρα πολύ σωστή παρέμβαση ε, με πολλά στοιχεία. Ο κύριος Τούρμες πρώτος. Πάρα πολύ ωραίο είναι που βλέπουμε διαφορετικές απόψεις από δύο σημαντικές ε, χώρες, ε, από τη Γερμανία και από την Πολωνία. Πριν μερικά χρόνια μου είπαν, αλλά δεν μπόρεσα να το ελέγξω, ότι υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Πολωνία. Παλιότερα, στην αρχή της αλλαγής ε, ε, καθεστώτος. Και μετά ε, η κυβέρνηση Γιαζίνσκι ε, ήρθε και δεν προχώρησε τη συμφωνία. Ιστορικά αποδεικνύεται αυτό. Γιατί ακούω ότι ο πρώτος North Stream δημιουργήθηκε γιατί η Πολωνία δεν ε, σεβάστηκε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει απέναντι στη Ρωσία. Αλλά είναι η ε, πραγματικότητα αυτή η επιχειρηματολογία ισχύει γιατί στη Γερμανία ακούγεται πολύ. Δεύτερον, αυτή αυτός ο νέος ε, αγωγός Νορβηγία, Δανία, Δανία, Πολωνία. Οικονομικά πώς μπορεί να λειτουργήσει 3 ή 13 BCM. Ποια είναι η άποψή σας. Και τελευταίο δουλεύω λίγο τώρα και τα θέματα της νοτιοανατολικής ε, Ευρώπης. Αλλά όλοι θέλουν να γίνουν ε, κόμβος ε, για το φυσικό αέριο. Η Βουλγαρία το θέλει. Η Ρουμανία είναι ίσως καλύτερα τοποθετημένη γιατί έχουν δικό τους, δικιά τους παραγωγή. Στην Ελλάδα όποιον και να ρωτήσει θα πει όχι, όχι, εμείς είμαστε το καλύτερο χάμπ. Αλλά τι γίνεται όταν ε, η παραγωγή ας πούμε, ή ε, ε, η κατανάλωση είναι μικρή. Εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε υγροποιημένο αέριο και χρειαζόμαστε τέτοια αγορά. Αλλά πώς μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω κάποιες χώρες. Ας πούμε η Σερβία κατά την άποψή μου που είναι μια χώρα που καταναλώνει πολύ αέριο, θα πρέπει και αυτή ε, να ενταχθεί σε αυτές τις διαδικασίες μαζί με τις άλλες βαλκανικές χώρες. Παρακαλώ πολύ συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε. Είναι ενδιαφέρον να δει ότι κανείς, ε, ο καθένας μάλλον προσπαθεί να ε, καλύψει τα δικά του συμφέροντα. Η Γερμανία θέλει να καλύψει ε, την ενεργειακή της προμήθεια και η Γαλλία το ίδιο βέβαια. Γιατί αν αύριο ας πούμε υπήρχε κάποια σύραξη ε, με την Πολωνία, με την Ρωσία. Ε, θα έπρεπε να έχουμε δυνατότητα διαφοροποίησης ε, της προμήθειας. Αυτό πάντως που διαπιστώνουμε είναι ότι πλέον δεν έχουμε ενεργειακή ασφάλεια. Πριν την είχαμε την ασφάλεια αυτή, γιατί δεν βλέπαμε από πολιτικό πρίσμα τις διαδικασίες. Δηλαδή ακόμα και αν δεν συμφωνούσαμε, που δεν συμφωνούσαμε ε, με την διακυβέρνηση της ε, Ρωσίας, ε, είχαμε διασφαλισμένη την προμήθεια ενέργειας. Τώρα όμως δεν συμβαίνει αυτό και εξ αυτού προκύπτει μια μεγάλη τροτότητα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας από πολιτική σκοπιά. Ε, εδώ πραγματικά δεν έχει τέλος επομένως αυτή η διαδικασία γιατί πρόκειται ε, για απόλυτα ε, υποκειμενικές απόψεις οι οποίες δεν οδηγούν καθόλου σε κοινή στρατηγική. Το είδαμε και με αυτά που λέτε για την Πολωνία, το βλέπουμε και με άλλες χώρες. Δεν υπάρχει κοινή πολιτική. Ε, θα ήθελα και εγώ μία πολύ σύντομη ερώτηση. Αναφερθήκατε ε, στην, στον ρόλο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι ώστε να, να υπάρχουν στο μέλλον ομοιόμορφοι κανόνες. Τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορεί η Κομισιόν να κάνει γι' αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ως προς τη συμφωνία μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας ε, δεν ε, καταλαβαίνω τι εννοείται επακριβώς. Υπήρχαν όμως δύο προγράμματα υποδομών που δεν ονοκληρώθηκαν. Υπήρχαν ε, πολλές παρεξηγήσεις και από πλευράς Πολωνίας και από πλευράς Ρωσίας και στη συνέχεια έγινε λόγος ε, για την μη χρησιμοποίηση της Ουκρανίας, να περάσουμε δηλαδή από τη Σλοβακία και την Πολωνία, να παρακάμψουμε την Ουκρανία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε και το ρόλο της Ουκρανίας στην ε, μετάβαση, στη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Όσον αφορά τον βαλτικό αγωγό και το ρόλο της ε, Νορβηγίας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι από πλευράς Πολωνίας να υπάρχει ένας ανεξάρτητος φορέας προμήθειας φυσικού αερίου για να υπάρχει μια ανταγωνιστική αγορά στην Πολωνία και στην περιφέρειά της. Και υπάρχει και το θέμα της ε, μείωσης της ε, ασφάλειας ε, ενέργειας, γιατί όπως ξέρετε θα σταματήσει να λειτουργεί ένας μεγάλος κόμβος, μια μονάδα, μια μεγάλη μονάδα στη Δανία, όπου υπάρχει και μια συνδεσιμότητα με τη Γερμανία σε σχέση με τους κόμβους και ε, που θα υπάρχουν ο καθένας θέλει να είναι κομβικό σημείο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχουν επιπλέον προμήθειες στην ευρύτερη περιφέρεια. Ακούσαμε ότι επενδύθηκαν 65 δις ευρώ στις υποδομές και μόνο ένα ε, απειροελάχιστο κομμάτι πήγε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, άρα δεν υπάρχει ανάπτυξη στις υπόδομες. Χρειαζόμαστε μια αγορά, αλλά μας ενδιαφέρουν και οι προμήθειες. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει στη ζήτηση, γιατί η Πολωνία δεν είναι μεγάλη αγορά ε, φυσικού αερίου, αλλά είναι κομβικό σημείο. Μετά υπήρξε και ένα σχόλιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ασφάλεια προμηθειών. Για μένα το βασικό ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για κοινούς στόχους, γιατί μπορούμε να ορίσουμε ε, ένα κοινό πλαίσιο, μια κοινή γλώσσα, για να σχεδιάσουμε και τα μέσα που χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ, δεν νομίζω ότι έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Και εγώ θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο Μπούζεκ, κάτι το οποίο είναι ασύνηθες, γιατί είναι η εισηγητής. Στην έκθεση αυτή κατανοώ απόλυτα και αυτά που είπατε στα Ιταλικά, και το οποίο με εκπλήσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε πολλή εργασία μπροστά μας, έχουμε δύο κανονισμούς, δύο ανακοινώσεις. Τώρα έχουμε αρχίσει με τις εργασίες μας και οι συζητήσεις θα μας βοηθούσαν ιδιαίτερα και για τις ε, μελλοντικές μας ε, φιλοδοξίες στην ε, Ήτρε σε σχέση με τις υποθέσεις εργασίας από την πρόταση της Κομισιόν πρόκειται για ένα αξιόπιστο, για μια αξιόπιστη αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Υπάρχει ασφάλεια προμηθειών, κάτι το οποίο έχει συνέπειες στην οικονομία μας. Θέλουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να έχουμε ένα αξιόπιστο πλαίσιο προμηθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για περιφέρειες ε, όπου θα υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, επιμερισμός δηλαδή ευθυνών και θα θέλαμε να να καλύψουμε τα κενά της νομοθεσίας μας. Αυτό είναι ύψης της σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει δηλαδή η ιδέα της αλληλεγγύης να μεταφραστεί σε ένα νομοθετικό έργο με πραγματικές ευθύνες. Αυτό θα ήταν μεγάλη υποστήριξη για το μέλλον και επίσης ως προς τις χώρες ε, προμηθευτές θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ως προς τις διεθνείς συμφωνίες. Εδώ μιλάμε για 36 χώρες, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει εμείς να διαχειριστούμε καλύτερα αυτό το πλαίσιο για να έχουμε χαμηλότερες τιμές και να είμαστε ένας δυνατός εταίρος στους προμηθευτές μας. Όλα βρίσκονται ενώπιον μας εμείς θα θέλαμε να φτάσουμε και σε διάβλους επίγουσας ανάγκης για προμήθεια φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην δημιουργηθούν άλλες κρίσεις στο μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να κηρύξουμε τη λήξη του σεμιναρίου μας, κάτι το οποίο ήταν πολύ, πολύ χρήσιμο σε όλους. Ευχαριστούμε και όλους τους ε, ομιλητές, λέει η κυρία Τόγια. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Αντιπρόεδρος Άντσεπ φτάνει όπου να είναι. Το περιμένουμε με χαρά. Και είναι το επόμενο θέμα στην ημερήσια διαταξή μας, αυτό της ανταλλαγής απόψε με τον κύριο Άντρους Άνσιπ. Αντιπρόεδρο Αρμόδιο για την ψηφιακή εσωτερική αγορά, διαρθρωτικός διάλογος, διαρθρωμένος διάλογος. Προχωρούμε. Λοιπόν, σε αυτό το διαρθρωμένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλώς ήρθατε. because you, you refused. <laughs> Well, uh, dear friends, let me remind all of you. Ε, υπενθυμίσω συνάδελφοι πως η Επιτροπή μας ε, ηγήθηκε αυτή της ε, πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ψήφισμα για την ψηφιακή αγορά που υιοθετήθηκε φέτος τον Ιανουάριο, από την οποία θα θα προκύψουν αρκετέ ε, αποφάσεις, απόφαση για το φάσμα, ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας, ε, αναθεώρηση τηλεπικοινωνιών που αναμένεται εντό λίγων μηνών και άλλες προτάσεις. Έχουμε πολλά λοιπόν να πούμε και υπενθυμίζω, συνάδελφοι, πως ο Αντιπρόεδρος Άνσιπ έχει προσκληθεί στο πλαίσιο αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου στην Επιτροπή μας, ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλους εμάς τους ευρωβουλευτές, και θα μας δώσει μια ενημέρωση για την ε, υλοποίηση πλευράς της Επιτροπής του Προγράμματος Εργασιών του 2016, αλλά και προοπτικές για το 2017 ταυτόχρονα. Τον έχουμε συναντήσει στη διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών πριν από δύο μήνες, όπου συζητήσαμε όλες τις πτυχές της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και τη δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είπε αυτή τη ενιαία. Έχουμε περίπου μια ώρα και δέκα λεπτά στη διάθεσή μας, αρκετός χρόνος και παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο να μας κάνει την παρουσίασή του. Εκφωνώντας το λόγο του. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Το προηγούμενο Μάιο, όταν ξεκίνησε η ψηφιακή ε, νέα αγορά, κάναμε δύο προτάσεις, εκ των οποίων η μία αφορούσε την ε, μεταφοριμότητα, αλλά και κανόνες συμβάσεων. Προτείναμε πιο εναρμονισμένους κανόνες για τις συμβάσεις. Το Φεβρουάριο Κάναμε μια πρόταση για τα 700 MHz που έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την ίδρυα αλλά και για μένα προσωπικά. Η Ολλανδική Προεδρία έκανε πολύ καλή δουλειά εν προκειμένου ε, σε αυτή την πρόταση δηλαδή για τα 700 MHz και αν θυμάστε είχαμε αποφασίσει να χωρίσουμε σε δύο τμήματα αυτά τα 700 MHz με τα ανώτερα φάσματα 694 δηλαδή έως 790 MHz για τους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και κάτω από τα 700 440 δηλαδή έως 694 MHz θα είναι το φάσμα διαθέσιμο για ψηφιακή ε, χερσαία τηλεόραση, ε, ασύρματα μικρόφωνα που ενδεχομένω χρησιμοποιούνται σε θέατρα και το καθεξής. Άρα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια στην υπόθεση αυτή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προβλεψιμότητα ε, και σαφήνεια, γιατί κανείς δεν γνωρίζει για πόσο διάστημα μπορεί να χρησιμοποιεί τις συχνότητες, χωρίς λοιπόν δυνατότητα πρόβλεψης δεν είναι και κανείς διατεθειμένος να προβεί σε επενδύσεις. Στόχος μας είναι λοιπόν να εξασφαλίσουμε αυτό το ανώτατο επίπεδο του φάσματος, το, το στρώμα του φάσματος για τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, γιατί βεβαίως θέλουμε και το, είναι υψηλή τεχνολογία, το ίντερνετ των πραγμάτων, και πρέπει ταυτόχρονα να παραμείνει διαθέσιμο και το χαμηλότερο στρώμα. Ε, η απόφαση θα είναι χρήσιμη και για τους παραδοσιακούς ε, τηλεοπτικούς σταθμούς που εκπέμπουν, θα γνωρίζουν για πόσο διάστημα θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές οι συχνότητες. Στο Συμβούλιο βέβαια κάποιες χώρες ζήτησαν μακρότερη περίοδο ε, προσαρμογής, όχι ως το 2020 αλλά το 2022 για την εφαρμογή. Ξέρουμε όλοι ότι στην Νότια Κορέα και την Ιαπωνία αρχίζουν να χρησιμοποιούν στοιχεία, σημαντικά κομμάτια του πακέτου των, ε, του 5G για τους Ολυμπιακούς που έχουν προγραμματιστεί για το 2018 και 2020. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε επίσης στόχο προδιαγραφών 5G για το 2020. Η Ericsson μας λέει ότι τουλάχιστον δύο πόλεις μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν μεγάλο τμήμα του 5G. από το 2018. Η Στοκχόλμη και το Ταλίν βεβαίως είναι αυτές οι πόλεις. Πρέπει να βιαστούμε λοιπόν. Και το θέμα δεν είναι πόσο γενναιόδωρο θα αποδειχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το μέλλον των χωρών μας, το μέλλον της Ευρώπης της ίδιας. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Πρέπει να αναλάβουμε ηγετική θέση στο παγκόσμιο σκηνικό. Βεβαίως, αντιλαμβανόμενοι ότι υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις στα κράτη-μέλη. Φερρυπίν, στην Φιλανδία, το φάσμα κάτω από τα 700 MHz δεν χρησιμοποιείται καν για την ε, χερσαία τηλεόραση και δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Άλλες χώρες όμως, η Ιταλία, έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για τη χερσαία τηλεόραση σε αυτό το φάσμα και άρα πρέπει να βρούμε λύσεις και για τις χώρες αυτές. Μπορούν να προκύψουν σημαντικές περιπλοκές λόγω της υψηλής χρήσης από τη χερσαία ψηφιακή τηλεόραση αυτού του ε, τμήματος του φάσματος. Περιπλοκές επίσης προκύπτουν σε σχέση με τα 700 MHz και σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι κατά τη Λοναλδική Προεδρία, τα κράτη-μέλη και κυρίως η Προεδρία έκαναν πολύ καλή δουλειά. και επέτρεψαν την εξασφάλιση μιας γενικής προσέγγισης στις 25 Μαΐου. Αναμένατε. Τον Απρίλιο ξεκινήσαμε το πακέτο για την ψηφιοποίηση βιομηχανίας για επικοινωνία νέφους. Τώρα έχουμε 700 δις συνολικά, 70 το χρόνο δηλαδή, από χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου, για την έρευνα την επιστημονική, η οποία σε διάφορους ε, εξυπηρετητές, σερβερ και νέφη, αναπτύσσεται, αλλά επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα, δεν μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα σε επίπεδο big data μεγάλων δεδομένων ε, ή δεδομένων μεγάλου όγκου που θα ε, χρειαζόταν για να αποδώσει καρπούς ε, η χρηματοδότηση από χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογουμένου και τα ερευνητικά κέντρα μας ζητούν ευρωπαϊκά επιστημονικά νέφη ή επιστημονικό νέφος, κάτι το οποίο έχουμε βάλει στο σχεδιασμό μας. Βεβαίως και προτεραιότητες ε, ως προς το σχεδιασμό ε, προδιαγραφών και προτύπων ψηφιακής τεχνολογίας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε εντοπίσει πέντε τομείς όπου θέλουμε να επιταχύνουμε τις δραστηριότητε μας. Το 5G πρώτα απ' όλα, το νέφος, το ίντερνετ των πραγμάτων, τα δεδομένα και η κυβερνοασφάλεια. Για να είμαι πολύ το η τυποποίηση θα πρέπει να παραμείνει σε μια διαδικασία εθελοντική και στην οποία θα ε, έχει τον πρωταρχικό ρόλο ο βιομηχανικό κλάδο. Ταυτόχρονα όμω αυτή η διαδικασία τη τυποποίηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τι εξελίξει, τι διαδικασίε αυτέ οι οποίες, όπως είπα, ε, για να ξεκινήσουν ορισμένες τάσεις χρησιμοποιούν χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Κορφανά, τα χρήματα του Ευρωπαίου Είναι όμως πολύ δύσκολο να παρεύουμε στο τομέα των ε, προτύπων και θα σας δώσω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πάνω από 600 διαφορετικές ε, προδιαγραφές και πρότυπα σχετικά με το ίντερνετ των πραγμάτων. και ίσως ε, ήδη πολλά από αυτά για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις να είναι πολύ δυσνόητα. Όλοι αυτοί οι οποίοι παράγουν ε, οικιακές συσκευές, παραδείγματι, και που επιτρέπουν την ε, διασύνδεση αυτών μέσω του διαδικτύου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να υπάρχει αυτή η αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας και άρα πρέπει να κατασταθεί ένα μικρό τσίπ μέσα σε ένα ψυγείο φερρυπίν μια ηλεκτρική σκούπα το κόστος του οποίου αυτή τη στιγμή είναι 50 ευρώ. Αν όμως μπορέσουμε να φτιάξουμε θέλουμε να έχουμε πρότυπα ανοιχτά, ευμετάβλητα, θα πρέπει το κόστος να μην είναι τόσο υψηλό για τον ε, καταναλωτή. Πρέπει να είναι στα 9 ευρώ το πολύ για, το κάθε, για την κάθε συσκευή. Είναι ζητήματα αγωνιστικότητας. Συναντήθηκα με, τον, ε, με την ε, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της IBM, την κυρία Ρομέτη, και συζητήσαμε για προσπάθειες κοινέ μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών για κοινέ ε, ανοιχτέ προδιαγραφές για το ίντερνετ των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν το σύνολο μέτρων για την ψηφιοποίηση έχει να κάνει και με το, νέα, με το νέο πρόγραμμα δράσης για την ε, ψηφιακή διακυβέρνηση. Θέλουμε μια βασική αρχή για τις επιχειρήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικά επιχειρησιακά μητρώα τα οποία δεν επικοινωνούν το ένα με το άλλο. Εάν κάποιο θέλει, παραδείγματι, να συνάψει μια συμφωνία εδώ, στο Βέλγιο, και δεν είναι Βέλγος, δεν μπορεί να γνωρίζει εάν η επιχείρηση, ο κύριος ή η κυρία που την εκπροσωπεί συγκεκριμένα, εκπροσωπεί την επιχείρηση αυτή. Και χρειάζεται για να έχει τα αποδεκτικά στοιχεία να τα δει σε χαρτί Άρα πρέπει ο καθένας να φέρνει ε, για κάθε σύμβαση τα αποδεικτικά ε, από την πατρίδα του και από το σχετικό Μητρό Επιχειρήσεων. Παράξενο ωστόσο τον 21ο αιώνα να πρέπει ακόμη να αποδεικνύουμε επί χάρτου την ιδιότητά μας και να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο να είναι δυνατόν η πληροφορία να διέρχεται τα σύνορα κατά τρόπο απρόσκοπτο. Την Τετάρτη λοιπόν. Θα κάνουμε την πρόταση για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ίσως δεν είναι τόσο θέμα της Επιτροπής σας, αλλά πάντως είναι μια πολύ σημαντική πρόταση. Και ασφαλώς αφορά και την ε, κατάργηση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού που είναι επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί 2% εκείνων οι οποίοι ήθελαν να αγοράσουν κάτι από μια άλλη χώρα με βάση τις τελευταίες έρευνες, δεν είχαν πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα, στον σχετικό ιστότοπο και 27% εκείνων που είχαν πρόσβαση στον ιστότοπο δεν μπορούσαν να ε, καταγραφούν, να εγγραφούν ως πελάτες και από αυτούς 32% ε, αυτοί που είχαν την τύχη και δεν, μπόρεσαν, δεν είχαν προβλήματα προς την εγγραφή, είχαν προβλήματα στην παράδοση. Και όσοι δεν είχαν προβλήματα στην παράδοση, δεν μπορούσαν να πληρώσουν. 26% εκείνων που δεν είχαν προβλήματα προς την παράδοση δεν μπορούσαν να πληρώσουν στο εξωτερικό. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μόνο 36,6% από όλους αυτούς τους ε, πολίτες που θέλησαν να αγοράσουν ε, αγαθό ή υπηρεσία από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπόρεσαν να το καταφέρουν. Αυτό δηλαδή σημαίνει εσωτερική αγορά. Αυτή είναι η δική μου ερώτηση. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν και πρέπει να τα λύσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επιβάλλουμε την υποχρέωση να πωλεί κανείς όπως σαν να ήταν ο Χωρί Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επιβληθεί υποχρεωτική παράδοση, ε, γιατί βεβαίω εκεί ε, θα ισχύει το εγχώριο, το οικείο, ε, εμπορικό δίκαιο. Δεν θα επιβάλλουμε βεβαίως τιμές για την αποστολή των προϊόντων, θα ισχύουν οι κατά περίπτωση τιμές, αλλά και σε αυτό θα πρέπει πιστεύω να παρέμβουμε γιατί είναι πολύ υψηλές πολλές φορές οι τιμές αποστολής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το κάνουμε αυτό και για το καλό των επιχειρήσεων και για το καλό των πελατών μας. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε και για τις ψηφιακές υπηρεσίες μέσω μας και σε αλλά και αυτό πάλι δεν, δεν αφορά τόσο πολύ στην Επιτροπή σας. Έχουμε πάντως να κάνουμε με την ε, ρύθμιση πλατφορμών επικοινωνίας και εδώ ασφαλώς θα εμπλακεί η δική Επιτροπή. Πλατφόρμες λοιπόν. Αποφασίσαμε να μην ακολουθήσουμε μια ε, εγκάρσια προσέγγιση, αλλά μια προσέγγιση αναπροϊόν ή ανα, πρόβλημα καλύτερα. Προβλήματα έχουμε ανάλογα με τις πλατφόρμες. Ε, κάποιοι παραδείγματι διαμαρτύρονται για απουσία διαφάνειες, Διαφάνειες όταν μιλούμε για ε, μηχανισμούς ε, αναζήτησης ως προς το πώς μπορούν να προβληθούν, πώς μπορεί κανείς να βρει την προβολή, αυτών των ε, σελίδων, γιατί πάντα εμφανίζονται οι πιο δεσπόζουσες επιχειρήσεις. Άλλοι βέβαια μας μιλούν για προβλήματα στην προστασία των δεδομένων, άλλοι μας μιλούν για προβλήματα φορολογικά. Ο κάθε φορέας λοιπόν που δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρεί τους ίδιους κανόνες και βεβαίως και εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες τεχνολογίες. Άλλους μπορεί να διαμαρτύρεται για το value gap, το κενό ε, ή το χάσμα στην αξία, μουσική επιτοπλίστων, που οργανώνουν ε, περιεχόμενο νόμιμο, αλλά που μπορεί να χρησιμοποιείται στη συνέχεια παράνομα και κάποιος τρίτος να κερδίζει, να αποκομίζει κέρδος από αυτό, χωρίς όμως να αποδίδει τίποτα. Και σε αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα υπάρχει πρόταση λοιπόν μέχρι το είναι Τετάρτη. Ξέρω ότι έχω ξαντλήσει το χρόνο μου. Ωστόσο, τον Ιούνιο θα κάνουμε την πρόταση για την κυβερνοασφάλεια ε, σε συμπράξει δημοσίου Με την ησυχία σας, λέει ο πρόεδρο, με την ησυχία σα χρόνο έχουμε. Επιταχύνω παρόλα αυτά, λέει ο κύριος Άνσιπ. Το Σεπτέμβριο. Πολύ σημαντική πρόταση και για την Επιτροπή σε σημαντική μεταρρύθμιση των κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες. Και στο επίκεντρο της πρότασης αυτής το φάσμα. Χρειάζεται βαθύτερο και πάλι εν προκειμένου θέλω να σημειώσω ότι είναι σαφές πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κοιτάει τι χρήματα αποκομίζουν τα κράτη-μέλη πολλώντας συχνότητες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα κράτη-μέλη θα αξιοποιήσουν τους φυσικούς τους πόρους και το φάσμα τους. Αλλά θέλουμε περισσότερο συντονισμό στο πεδίο αυτό. Μπορούμε, Φερρυπή, να οροματιζόμαστε συνδεδεμένα αυτοκίνητα που θα περνούν ε, τα σύνορα ε, αλλά αυτό χωρίς ε, βαθύτερο συντονισμό δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ, θα παραμείνει στο πεδίο του, φανταστικού. Χρειάζεται λοιπόν να συντονιστεί ο, ε, ο χρονισμός αυτών των δημοπρασιών φάσματος, πρέπει να συντονιστεί η διάρκεια των αδειών και από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι καλύτερο να υπάρχει μεγαλύτερη διάρκεια για τις αδείες στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι απεριόριστες χρονικά μάλιστα Κάποιοι πρότειναν 25 χρόνια. 25 χρόνια ασφαλώς είναι καλύτερα από τα 5, γιατί μια πολύ σύντομη χρονική περίοδος δεν θα επιτρέψει κανέναν να προχωρήσει σε πραγματικές επενδύσεις. Επίσης, συντονίζουμε την κάλυψη των ε, συχνοτήτων γιατί η εικόνα είναι πολύ διαφορετική αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως είπα μπορεί να οραματιζόμαστε συνδεδεμένα αυτοκίνητα και γι' αυτό χρειάζεται βαθύτερο τονισμός και ως προς την κάλυψη των δρόμων. Συντονισμός λοιπόν, αλλά και επενδύσεις, επενδύσεις στην Ήπεθρο και το καθεξής. Και για το τελευταίο μου ε, σημείο, πρόταση για την προστασία των δεδομένων. αλλά και μια γενική αναθεώρηση που να αναφέρω τον Ιούνιο Από τις 15 Ιουνίου του 2017 έχουμε καταργήσει βεβαίως ε, το κόστος περιαγωγής, θα καταργηθεί το κόστος περιαγωγής, αλλά πρέπει και στις ε, τιμές της χονδρικής να βρούμε κάποια λύση. Και οι τελευταίες προτάσεις αφορούν την οδηγία για την, ηλεκτρονική, για την προστασία του ιδιωτικού χώρου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, προστασία των ε, δικαιωμάτων πνευματικής διοκτησίας και τη σχετική οδηγία για την επιβολή αυτής. Αυτά. Ξέρω ότι δεν ήμουν σύντομος και στο συγγνώμη. Πολύ ωραία. Ακούσαμε λοιπόν μια σειρά από από εσά και θα ξεκινήσουμε τώρα τις ερωτήσεις, σχόλια, τις παρατηρήσεις εξ ονόματος του ΕΛΚΑ ο κύριος Μπόνι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας, για τις πληροφορίες που μας δώσατε, καθώς επίσης και αυτήν την ε, ολιστική άποψη που μας δώσατε για τα ψηφιακά ζητήματα. Πριν από ένα μισή χρόνο ξεκίνησε η διαδικασία για την ενιαία ψηφιακή αγορά και νομίζω ότι δεν προχωράμε πολύ γρήγορα, αλλά τουλάχιστον προχωράμε με αποφασιστικότητα. Και αυτή η αποφασιστικότητα είναι ακριβώς σημαντική, διότι θα μας δώσει την δυνατότητα να λάβουμε υπόψη μας ε, όλα τα στοιχεία που αφορούν το πρόβλημα. Εγώ θα εστιάσω την ε, παρουσίασή μου σε ορισμένα στοιχεία. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι να κατανοήσουμε ότι για να επιτευχθεί η οικοδόμηση της ψηφιακής αγοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεπεράσουμε ε, κάποιες, να καλύψουμε κάποιες τεχνικές προϋποθέσεις. Αναφερθήκατε σε ορισμένες από αυτές, ας πούμε την τυποποίηση. Ερώτηση λοιπόν. Με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην ε, ανάμεσα σε ένα ε, ε, ε, βιομηχανικό μοντέλο τυποποίηση σε εθελοντική βάση, ενώ ταυτόχρονα να προωθήσουμε τις διαδικασίες τυποποίησης, να προωθήσουμε τις διαδικασίες και τα τεχνικά πρότυπα όσον αφορά και το ίντερνετ των πραγμάτων κλπ όσον αφορά την διαλειτουργικότητα και όσον αφορά και την, ε, ε, την ηλεκτρονική ταυτότητα αλλά και την πρόθεση μεταξύ των κρατών μελών ταυτόσιμων λύσεων. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Έχουμε πολλές παρόμοιες ιδέες όσον αφορά την πιστοποίηση και την ταυτοποίηση. Αλλά από την άλλη πλευρά φοβάμαι ότι στα κράτη-μέλη δεν ε, ε, θα είναι όλα έτοιμα ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, έτσι ώστε να ακολουθήσουν όλοι την ίδια πορεία. Τρίτο, ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο και η μορφή του. Βλέπω ότι η Κομισιόν προσανατολίζεται όχι μόνο και απλά σε ισχυρότερη ρύθμιση, γιατί αυτό είναι κάτι καλό, αλλά βλέπω ότι θέλει να προτείνει και κάποια στοιχεία τα οποία σχετίζονται ε, με τα PPPs ε, ή κάποιες προτάσεις ε, οι οποίες θα σχετίζονται ας πούμε με την, τις βέλτιστες πρακτικές και τον κώδικα δεοντολογίας. Όλα αυτά είναι καλά, γιατί είναι καλό να υπάρχει soft law, αλλά παρόλα αυτά ε, θα πρέπει ας πούμε, για θέματα όπως είναι ο ανταγωνισμός, η τεχνολογία και η καινοτομία, θα πρέπει να διέπονται από ισχυρή νομοθεσία. Το τελευταίο στοιχείο μου αφορά τις πλατφόρμες. Τα Υπουργεία κάποιων Ευρωπαϊκών χωρών στο Συμβούλιο Ενέργειας, Ανταγωνισμού κλπ. υπέβαλαν ε, μια επιστολή και σε εσά και στην Προεδρία αναφέροντας κάποιες ε, προτάσεις σχετικά ε, με την ενιαία αγορά η οποία θα πρέπει να γίνει ε, ψηφιακή ε, αποφεύγοντας όμως οποιαδήποτε επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια λοιπόν για τις πλατφόρμες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπεθ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτρεπε. Φέτος ολοκληρώνεται ένας χρόνος μετά την παρουσίαση της ε, στρατηγικής για την ψηφιακή αγορά ε, που αποτέλεσε μία από τις προτεραιότητες ε, της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη το Κοινοβούλιο έχει εκφραστεί για τη στρατηγική αυτή μέσω έκθεσης δια της οποίας εμείς ζητούσαμε να προωθηθεί η ψηφιοποίηση αλλά να αντιμετωπιστούν και κάποιοι σαφείς κίνδυνοι ε, και όσον αφορά δηλαδή τις ελλείψεις μεταξύ και το, όσον αφορά το μεγάλωμα του χάσματος του ψηφιακού και μεταξύ γενεών και μεταξύ ε, περιφερειών. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο αναφερθήκαμε, στο οποίο αναφερθήκαμε είναι η προστασία ε, των ε, επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων, γιατί αυτά δεν έχουν υπογραμμιστεί αρκετά. Επίσης, η Κομισιόν θα πρέπει να μας δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τις προτεραιότητες, τις οποίες στην ανακοίνωσή της ανέφερε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία θα πρέπει να δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Κομισιόν. Έχουμε την εντύπωση πάντως ότι κάποιες από τις προτάσεις ε, δεν, ε, έχουν, δεν είναι πολύ συγκεκριμένες. Ε, ας πούμε, όπως και η δέσμη για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας που είναι σημαντικότατη ε, θεμελιώδη σημασία για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ε, αναφέρεται η προστασία των ε, εργαζόμενων σε αυτούς τους τομείς ενώ τελικά αναφέρεται μονάχα κάτι πολύ πιο απλό δηλαδή ο διάλογος μεταξύ της βιομηχανίας και των κοινωνικών εταίρων. Επίσης ε, το ε, θέμα των επενδύσεων που ξεπερνούν τα 5 δις ε, που αποτελούν βεβαίως ένα μεγάλο ευρύ πλαίσιο όπου όμως δεν αναφέρεται καθόλου σε συγκεκριμένα και επιμέρους απτά προγράμματα. Επίσης το θέμα του νέφους και εδώ θα γίνεται λόγος ε, για 6,7 ε, δις επενδύσεων, εκ των οποίων τα μισά περίπου ε, θα αφορούσαν επενδύσεις ιδιωτικές. Ε, αλλά δεν ε, τίθεται ε, επιτάπητος το θέμα της αναθεώρησης του geoblocking, των πλατφορμών του διαδικτύου και άλλων στοιχείων. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά να προσπαθήσουμε έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες και η Ευρώπη στο σύνολό της να μπορέσει να ε, ε, εκμεταλλευτεί το ψηφιακό περίπτωμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Δελκαστίγιο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντιπρόεδρε. Πριν από ένα χρόνο η Κομισιόν ε, παρουσίασε ένα πρόγραμμα αναφερόμενο αναφερόμενοι στην ε, ε, ψηφιακή αγορά και θεωρώντας ότι είναι ε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εσείς είσαστε επικεφαλής αυτής της διαδικασίας. 18 μήνες έχουν περάσει και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Κομισιόν έχει ξεκινήσει ήδη να παραδίδει με την έννοια ότι βλέπουμε ε, αρκετές πρωτοβουλίες, άλλες νομοθετικές και άλλες όχι. Βλέποντας όμως όλα αυτά τα κείμενα, η πρώτη μου εντύπωση, η εντύπωση είναι ότι δεν πρέπει να χάσουμε καθόλου χρόνο, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2018 και να, να φτάσουμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου ε, θα έχουμε πάρει όλες τις σημαντικές ε, αποφάσεις ε, σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα 16 σημεία δράσης τα οποία έχετε παρουσιάσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. γιατί όντως ε, έχουμε το θέμα της, ε, του ε, e-commerce, έχουμε το geoblocking, είχαμε την φορητότητα, ένα σωρό κείμενα, αλλά λέω δεν έχουμε καθόλου χρόνο για χάσιμο, γιατί πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι στο τέλος ε, της ε, θητείας ε, θα μπορέσουμε να έχουμε φτάσει και να έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη σειρά των προτάσεων με την οποία συμφώνησε το Κοινοβούλιο και θα πρέπει το 2019 θα πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτή η αγορά που είναι η ενιαία ψηφιακή αγορά ε, που αποτελείται αυτή τη στιγμή από 28 κράτη ε, να μην υφίσταται πια, να είναι μια πραγματικά ενιαία αγορά. Ε, νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε τα μάλλον να συμβάλλουμε στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ. Roaming. Μιλάμε για μια Ευρώπη που θα απομακρυνθεί από το roaming το, του χρόνου, μέχρι του χρόνου. Γκρίφιν, ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο ανταγωνισμός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Θα πρέπει οι καταναλωτές να είναι στην καρδιά του προβλήματος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια μέτρα θα λάβετε έτσι ώστε τα δικαιώματα των καταναλωτών ε, να είναι στην καρδιά των μελλοντικών μέτρων. Υπάρχει ψηφιακό χάσμα σε σχέση με αυτούς που έχουν πρόσβαση στην τελευταία τεχνολογία και εκείνους που δεν την έχουν. Τη στιγμή που υπάρχει επιγραμμική επικοινωνία, υπάρχουν και αυτοί που γνωρίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, ιδιαίτερα στον τομέα της ε, ηλεκτρονικής υγείας και των μικρών επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν το ευρυζωνικό να είναι της τάξης ε, των 10 ε, MB ανά γιατί τα 30 MB ήταν ε, ο στόχος, αλλά μόνο το 40% των οικοκυριών έχει αυτή την ταχύτητα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μόνο το, ότι το 8% των ε, επιχειρήσεων και των πολιτών δεν έχουν πρόσβαση στο ευρυζωνικό με αυτή την ταχύτητα. Πώς θα λάβετε υπόψη όλες τις αγροτικές περιοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο ευρυζωνικό όπως ισχύει στα αστικά κέντρα. Ένα 40% των εργαζομένων ε, δεν έχουν ψηφιακά προσόντα. Πώς ε, προβάλλεται το θέμα με τις επιχειρήσεις και τα συνδικάτα έτσι ώστε οι εργαζόμενοι αλλά και οι νέοι να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να έχουν αξιοπρεπή εργασία σε ένα ψηφιακό κόσμο. Ρούμπιχ. Ευχαριστώ Πρόεδρο γιατί ε, θα ήθελα να πω ότι για μένα αυτό που έχει σημασία ιδιαίτερα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα ευρυζωνικό ώστε να μπορούμε να κινηθούμε και πέρα των σύνορων. Το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη θα πρέπει να βοηθήσει στη χρήση των οπτικών ινών στις τηλεπικοινωνίες από το 2018 αν ε, χρησιμοποιηθεί, γίνει σωστή χρήση και έχετε δίκιο ε, ότι τα χρήματα των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας ε, ανήκουν στους πολίτες. Δηλαδή μιλάμε για κεφάλαιο της ΕΤΕ. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα είχαμε μία ανάπτυξη των υποδομών Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να προωθήσει σχέδια και προγράμματα και οι Υπουργοί Οικονομικών θα βοηθούσαν και την ΕΤΕ. Θα υπήρχε δηλαδή μία ανάδραση. Θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε αυτό τον όγκο χρημάτων και επενδύσεων. Και αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη μία συνεχή ε, κινητικότητα και ταχύτητα για να δούμε ποια είναι η αποδοτικότητα σε σχέση με την μείωση του άχθου στο περιβάλλον. Και αυτό βεβαίω φαίνεται και μέσα από το Ιντερνετ. Θα πρέπει να δούμε ωστόσο τι είδου στατιστικέ ε, μπορούμε να έχουμε ώστε να, προσφέρεται ώστε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια σταθερή ταχύτητα, σε ποια κράτη είναι σταθερή ταχύτητα, χωρίς δηλαδή επιβραδύνσεις ή επιταχύνσεις ε, ε, των δεδομένων. Ευχαριστώ, Ζουρίνιο. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω και εγώ. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για τον πρώτο χρόνο της ε, ψηφιακής ατζέντας, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον και τι δεν πήγε καλά στο παρελθόν. Εμείς δεν κινηθήκαμε τάχιστα και δεν επικοινωνούμε ολοκληρωμένα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη αυτά τα δύο μηνύματα. Είπατε ότι όποιος θέλει να λειτουργήσει σε αυτή την εξαιρετική αγορά θα πρέπει να δεχτεί τους κανόνες μας, αλλά οι κανόνες μας θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. Να λάβουμε υπόψη δηλαδή το νέο πλαίσιο της ψηφιακής αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν η κοινή μας γνώμη, οι πολίτες να είναι σύμμαχοι για να ορίσουμε και τους ε, ρυθμιστές, να τους πιέσουμε έτσι ώστε αυτή να είναι μία κατά προτεραιότητα ατζέντα. Πιστεύω λοιπόν ότι όταν η Κομισιόν παρουσιάσει τη δεύτερη φάση του πακέτου θα πρέπει να υπάρξει μία ανακοίνωση όχι μόνο τεχνικής ήθης να μιλήσουμε για τον νέφος, για τα πνευματικά δικαιώματα και ούτω καθεξής. Θα πρέπει όμως να υπάρχει μια ολοκληρωμένη ανακοίνωση. Γιατί μιλάμε για ένα στοιχείο που θα κάνει διαφορά για την ποιότητα της ζωής των πολιτών και πιστεύουμε και αναμένουμε το, τον πυρήνα των προτάσεων. Η κυρία Κραήρ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ Επίτροπε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας. Δεν θα όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Θεωρώ ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την ουσία, με την πεμπτουσία της πολιτικής μας για τα επόμενα χρόνια και έχει να κάνει βέβαια και με τις υποδομές και με την νομοθεσία ασφαλώς. Ε, δεν ε, ήθελα λοιπόν ε, να αναπτύξω όλα αυτά, αλλά έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Είπατε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με την πολιτική στη με, τη... με το φάσμα και έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση σε σχέση με την χρήση φάσματος από τις ε, εκδηλώσεις και τους οργανωτές εκδηλώσεων. Είναι γνωστό το πρόβλημα. Η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής μόνο πει ότι για διάφορες εκδηλώσεις, ε, θεατρικές παραστάσεις, ε, συναυλίες και διασκέψεις και ό,τι άλλο χρειάζονται ρυθμίσεις που μπορεί να είναι και ευρωπαϊκές αλλά και εθνικές. Ερωτώ λοιπόν, γιατί έχουμε συστήσει επανειλημμένως, έχετε συγκεκριμένα σχέδια για την κάλυψη των αναγκών που είναι ε, μικρές γιατί αφορούν ένα μικρό κομμάτι της αγοράς αυτών των διοργανωτών αλλά που σε τελευταία ανάλυση ε, εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε μια καλή λύση θα υποστούν ε, δυσμενή μεταχείριση δεδομένου ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη ισχύ σε σχέση με άλλους παρόχους. Σας ευχαριστώ Σάντε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σε ορισμένες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλάμε για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών. Ο καλύτερος τρόπος είναι να υπάρχει ευρυζωνικό παντού σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια και ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό. Θα πρέπει να ορίσουμε νέους τρόπους εργασίας και ιδιαίτερα τηλεεργασίας, ιδιαίτερα στον αγροτικό κόσμο που βρίσκεται σε απομακρυσμένες περιοχές χρειάζονται το ευρυζωνικό για να μπορέσουν να προωθήσουν αυτές τις ε, πρακτικές για να υπάρχει και τηλεκατάρτιση και τηλεεκπαίδευση. Δύο είναι οι ερωτήσεις. Ποιες είναι οι λύσεις ε, για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και τι χρηματοδότηση μπορεί να προβλεφθεί. Κύριε Επίτροπε, Μιλήσατε ε, για συνδεσιμότητα, μιλήσατε για 600, 600 διαφορετικά πρότυπα και επίσης ε, μιλήσατε για ε, ε, οικιακό εξοπλισμό που αντί για 60 ευρώ θα μπορούσε να στοιχίζει Μιλάμε λοιπόν για τσιπάκια τα οποία θα μπορούσαν να, το κόστος το οποίο θα μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί στο 1 ευρώ. Αυτό μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να υπάρξει μία σωστή επεξήγηση και διάφρωση έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη αυτά τα τσιπάκια των ε, ηλεκτρικών συσκευών. Ας ε, δούμε αυτό το θέμα του ψηφιακού για να δούμε τι κάνει ακριβώς η Ευρώπη για να υπάρξει ε, μία, ένα πραγματικό οικοδόμημα και να μην ε, δώσουμε δίκαιο σε αυτούς που καταγγέλουν και κατηγορούν την Ευρώπη. Υπάρχουν ε, άλλοι που θα ήθελαν να ζητήσουν το λόγο. Θα ήθελα και εγώ, κύριε Επίτροπε, να προσθέσω μία ερώτηση σε σχέση με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιήσουμε αυτό το φάσμα των 700. Ε, Θεωρείτε από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει. Φαντάζομαι και στη δική σας χώρα ισχύει το ίδιο. Ένα άλλο ε, αμφίσιμο ζήτημα έγκυται στο εξής. Τι απάντηση θα μπορούσαμε να δώσουμε στο θέμα της ε, ε, πιθανότητας επιρροής του Wi-Fi, του ασύρματου δικτύου στην υγεία μας. Τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ευρυζωνικό υψηλής ε, ταχύτητας μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο ευρέως. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες, όλες αυτές τις ερωτήσεις τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τις στρατηγικές επενδύσεις. Καταρχάς, νομίζω για μένα είναι μια πολύ καλή πρόταση, πολύ καλή ιδέα. Στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε τις να προσελκύσουμε τις, τις επενδύσεις ώστε να αποδώσουν στο δυνατόν καλύτερα τα χρήματα που θα διαθέσει ο Ευρωπαίο φορολογούμενο και βέβαια να είναι το περιβάλλον στο δυνατόν καλύτερο για τι επιδοτικέ επενδύσει. Φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο τώρα δουλεύει. Και θα μπορούσα να σα πω κι άλλα. Το πρόβλημα να μην επισκεφθούμε την Αφρική, όπου κάναμε συζητήσει με την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, η οποία επίσης έδειξε ενδιαφέρον να αρχίσει να χρησιμοποιεί αντίστοιχο μοντέλο. Αν λοιπόν μπορέσουμε να προσελκύσουμε δυτικέ επενδύσεις, θα πει ότι θα δουλέψει το μοντέλο αυτό, το έργο αυτό. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρούμε λύσεις για επενδύσεις και σε άλλους τομείς. Για το Wi-Fi. Είδα κάποια άρθρα. Το οποίο όμω δεν στήριζαν σε κάποια έρευνα σχετικά με τις συνέπειες στην υγεία. Φήμες. Μόνο. Όχι επιστημονικά στοιχεία όμως. Και βέβαια πρέπει να προσέχουμε πολύ σε σχέση με τα επίπεδα των εκπομπών πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή και στο ίντερνετ των πραγμάτων. Δεν μπορούμε να εκτιθέμεθα σε μικροκύματα, παραδείγματι, μαζικά. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε μια σειρά από τεχνολογίες με μεγάλη προσοχή. Και το καλώδιο. Δεν είναι κακό. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να συντονίσουμε τις ε, δραστηριότητες μας για σε διαπραγματεύσεις με τους εταίρους ε, γείτονες ε, σε σχέση ειδικά με τα 400 MHz γιατί υπάρχουν με τα 700 MHz γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν τα 700 MHz για στρατιωτικούς σκοπούς. Και αυτό είναι στα πρόκληση βέβαια. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτές τις ε, συχνότητες για τους παρόχους όταν είναι πολύ ισχυρά τα σήματα από τις γειτονικές τους χώρες μέσα στο ίδιο φάσμα, στο ίδιο μικρό σχήματος. Ε, θα πρέπει να βρούμε λοιπόν μαζί τους μια λύση. Μέσα στον χρόνο έχουμε κάνει προτάσεις, αλλά έχουμε λάβει και κάποιες αποφάσεις, μπορώ να πω. Έχουμε αυτή την ε, Ευρώπη χωρίς κόστος περιαγωγής που την προετοιμάζαμε τόσα χρόνια. Και θέλω να σας θυμίσω από πού ξεκινήσαμε. Πού βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν. 5 συν 5 συν 5 ήταν η πρόταση. 5 λεπτά τηλεφώνημα πέντε ε, μηνύματα κινητά και 5 μεγαμπάιτ σε τιμές όσο και στην εγχώρια αγορά. Και φτάσαμε στο μηδέν. Καταφέραμε να καταργήσουμε ο, εντελώς το κόστος περιεγωγής. από τις 15 Ιουνίου του 2017 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλη μια φορά, σας παρακαλώ, να ασχοληθείτε πολύ εντατικά με την πρόταση αυτή. Ενώψε της 15 η Ιουνίου. για την αναθεώρηση της χίδιν παροχής. Και βέβαια η οδηγία μης για την ασφάλεια του δικτύου έχει πολύ μεγάλη σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη. Φυσικά δεν είναι δική μου θέση να, δεν είμαι σε θέση να δώσω υποδείξει στο κοινοβούλιο, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει και το κοινοβούλιο να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Και η μεταρρύθμιση του ίντερνετ των πραγμάτων έχει τεράστια σημασία για το μέλλον μας. Κύριε Μπόνη, θα συμφωνήσω μέσα ότι πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς, γιατί ο χρόνος τελειώνει. Όλοι μας όμως πρέπει και να αντιληφθούμε πως πρέπει να δώσουμε και τον χρόνο για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Η αποτελεσματική λοιπόν λήψη αποφάσεων, εάν δεν ακολουθεί τους κανόνες της δημοκρατίας, αν δεν γίνεται με δημοκρατικό τρόπο, δεν μπορεί να είναι τόσο καλή. Επίσης, σωστή ισορροπία μεταξύ μιας ε, προσέγγισης εθελοντικής ή αυτοδέσμευσης και επιβολής κανόνων. Κάποιοι διαμαρτύρονται για την επιβολή προτύπων. Θεωρούν δηλαδή ότι τα πρότυπα είναι κάτι το κακό. Έναντι της χρήσης του ε, λογισμικού ανοιχτής πηγής. Αν όμως εμείς συμφωνήσουμε ότι θα συναντηθούμε κάπου, δίνουμε ένα ραντεβού, αλλά δεν λέμε ακριβώς πού είναι αυτό το κάπου, Μπορεί ο ένας μας να αρχίσει να πηγαίνει προς τη μία κατεύθυνση και ο άλλος προς την άλλη. Και να μην συναντηθούμε ποτέ. Για μένα λοιπόν η τυποποίηση έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το σημείο συνάντησης. Ανοιχτά πρότυπα, θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λογισμικό ανοιχτή πηγής, αν υπάρχει ανάγκη. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα-δύο τουβλάκια, βεβαίω θα το πράξουμε. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε στο σημείο συνάντησης. για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες που συζητήθηκαν μάλιστα προσφατά σε μια ε, διάσκεψη που ήμουν και εγώ σήμερα και ο κύριος Μπόνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ο κανονισμός Άιντας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί τη βάση για τόσες τόσες πολλές ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρονται από το δημόσιο των κρατών μας ή από τις δυτικές επιχειρήσεις. Θα προχωρήσουμε λοιπόν. Ρυθμιστικό πλαίσιο. Ναι. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον και, τον και βέβαια να παραμείνουν εθνικές οι εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές ανεξάρτητες, αλλά πρέπει ταυτόχρονα και το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο να αρχίσει να διαμορφώνεται. Θα τα εξετάσουμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε με την αναθεώρηση. Χρονοδιάγραμμα για φέτος. Είναι πολύ πυκνό και σκληρό. Πάντα μπορούμε να λέμε πως χρειάζονται περισσότερες φιλοδοξίες και εγώ θέλω να είμαι πιο φιλόδοξος. Ο στόχος μου όμως δεν είναι να κάνω τις πιο φιλόδοξες προτάσεις του κόσμου. Εάν αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν. Τι στόχο θα έχουμε εγώ λοιπόν θέλω να φτάσω σε συγκεκριμένους στόχους και να είμαι βέβαιος πως θα είναι δυνατή η ε, ανέβρεση συνένεσης μεταξύ 100 μελών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χωρίς να θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με κανέναν θα θέλω να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψηφιακό ζήτημα έδειξε Μεγάλη φιλοδοξία. Συμφωνώ με την κυρία Πιλάρδη Ούτε λεπτό δεν πρέπει να χαθεί. Ο χρόνος τρέχει. Και βέβαια έχουμε και την πρόταση για τη στρατηγική για δεξιότητες όπου ξέρουμε πολύ καλά ότι σε 90% των θέσεων εργασία που ανοίγουν απαιτούνται κάποιου τύπου έστω ψηφιακέ δεξιότητε. Για μένα λοιπόν αυτή η στρατηγική θα έχει ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες. καταναλωτές και ψηφιακό χάσμα. Είναι όντως μεγάλη πρόκληση. Γιατί και στις χώρες που έχουν ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ψηφιακά θέματα παραμένει το ψηφιακό χάσμα. Το ψηφιακό χάσμα είναι αυτό που υπάρχει μεταξύ εκείνου που μένει στην Ήπεθρο και εκείνου που μένει σε ένα κέντρο πόλης, μεταξύ του πιο ηλικιωμένου και του νεότερου. Αλλά ψηφιακό χάσμα υπάρχει και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι όλα αυτά θέματα που θα πρέπει βεβαίως να αντιμετωπίσουμε ήδη η πρόσβαση στο ίντερνετ πρέπει να είναι πιστεύω ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα γιατί αφορά την πρόσβαση στην πληροφορία. Και αυτό όχι για ένα χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά για την πραγματικότητα πρέπει να εντάσσεται στα θεμελιώδη δικαιώματα. Για τις περιοχές της Πέθρου πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ιδιαίτερες λύσεις για την ναι, έπιστευμα στον ανταγωνισμό εάν ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, πιστεύω ότι θα υπάρχει καλό περιβάλλον και για την καινοτομία και για τις επενδύσεις. Κάποιοι πάροχοι βέβαια λένε ότι είναι πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός, δεν έχουμε οικονομική επιφάνεια πλέον για επενδύσεις. Βλέπουμε όμως από την πραγματικότητα ότι πραγματοποιούνται, ε, υλοποιείται καινοτομία, προχωρεί η καινοτομία και όταν υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός αυτός κινητοποιεί τον επενδυτή όταν είναι πραγματικά σκληρός. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές όπου η πυκνότητα πληθυσμού είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι στα μεγαλύτερα κέντρα δεν είναι τόσο ελκυστικό το περιβάλλον για, τον, ε, για την ιδιωτική επένδυση. Και πρέπει και αυτό το περιβάλλον να το καταστήσουμε ε, ελκυστικό για τις ιδιωτικές επενδύσεις, γιατί όπως είπα αφορά βέβαια τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά αυτό ξέρετε και η οικονομία μας, η γεωργία μας. Να προσφέρουμε πρόσβαση για την ευρυζωνικότητα και στις περιοχές υπαίθρου. Τα τελευταία 20 χρόνια ξέρουμε ότι οι τιμές παραγωγικότητας στο γεωργικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν ε, γεωμετρικά. Η Εστονία που σας ανέφερα και νωρίτερα ως παράδειγμα πριν από 25 χρόνια είχε 3,5 τόνους γάλα παραγωγή ανά αγελάδα το χρόνο κατά μέσο ώρα. Τώρα είναι στα 5,2, στους 5,2 τόνους. Πώς το καταφέρει είναι ένα παράδειγμα της οικονομίας της βασιζόμενης στη γνώση. Χάρη στο ίντερνετ τα καταφέραν. Γιατί είναι μηχανήματα αυτά τα οποία αρμέγουν τις αγελάδες πια. Και αυτά τα οποία φροντίζουν για την ζωοτροφή τους κτλ. Με βάση την οικονομία της γνώσης. Και έτσι μπόρεσαν από τους 3,5 τόνους τον χρόνο να φτάσουν στους 8,2 τόνους γάλα παραγωγή Αφορά λοιπόν και το γεωργικό μας τομέα. Στην Ιταλία μαθαίνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείται το ίντερνετ και για την παραγωγή καλού κρασιού. Το ίντερνετ λοιπόν, μια προσέγγιση στηριζόμενη στη γνώση, έχει μεγάλη σημασία σε κάθε τομέα. Τι έχουμε υπόψη λοιπόν για την Ήπεθρο. Νέα μοντέλα παραχωρήσω, Προστασία σε εκείνους που είναι διτεθειμένοι να κάνουν πρώτη την επένδυση. Στη Γερμανία, παραδείγματι, υπάρχει μια πόλη όπου και ο Δήμος αλλά και ένας ιδιώτης επενδυτής αποφάσισαν να επενδύσουν σημαντικό ποσό στην ευρυζωνικότητα. Και όταν έχει γίνει αυτή η επένδυση, α, τους ακολούθησε και άλλη μια εταιρεία. Και έκανε και εκείνη επενδύσεις. Πρέπει να εξασφαλιστεί λοιπόν ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στον κάθε φορέα και να εξασφαλιστεί η προστασία, ένα περιβάλλον τέλο πάντων κατάλληλο ώστε να προστατευθεί εκείνος ο οποίος πρώτος κάνει την κίνηση. Σκεφτόμαστε και για κοινέ ε, επενδύσεις, ε, για προστασία λοιπόν των επενδύσεων στην Ήπεθρο και ο στόχος μας είναι να καλύψουμε ολόκληρη την Ήπεθρο με ίντερνετ υψηλής ταχύτητας. Οι Υπουργοί βέβαια των οικονομικών που βάζουν και τα ανώτατα όρια στη χρηματοδότηση, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους. Πρέπει να τους εξηγήσουμε και τι είναι το φάσμα και τι είναι οι συχνότητες και είμαι βέβαιος ότι στις χώρες εκείνες όπου οι κυβερνήσεις δεν επιδιώκουν μόνο τη μέγιστη οικονομία σε πόρους, και την, ε, το μέγιστο κέρδος από την πώληση των συχνοτήτων. Πιστεύω ότι αυτές οι χώρες που δεν επιδιώκουν το μέγιστο κέρδος από την πώληση των συχνοτήτων κάνουν μεγάλο σφάλμα. Και είναι σε άλλες κυβερνήσεις οι οποίες κοιτούν πιο μακρόπνοα και ορίζουν συγκεκριμένους όρους, προδιαγραφές, προϋποθέσεις και χρονικά όρια για την αξιοποίηση του φάσματος θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα και έσοδα καθώς οι οικονομίες τους θα αναπτυχθούν ταχύτερα χάρη στη νέα τεχνολογία που θα είναι διαθέσιμη. Είδαμε ήδη τον αντίκτυπο του 4G μεταξύ, και τις διαφορές των αντίκτυπων μεταξύ φορών κρατών. Ελπίζω πως όταν έρθει η ώρα για το 5G θα έχουν ορίσει όλες οι χώρες συγκεκριμένου όρους και θα ζητήσουν αμέσως το υψηλότερο τίμημα, αλλά θα κοιτάξουν πιο μακροπρόθεσμα, ώστε ο καθένας εν τέλει να βγει κερδισμένος. Ευελιξία, ναι. Πρέπει να υπάρξει ευελιξία όταν μιλούμε για 700 MHz. Το είπα ήδη στην αρχή οι χώρες μας, τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε διαφορετικές ε, καταστάσεις και σε ορισμένες χώρες όπως είπαμε δεν αξιοποιούνται, δεν χρησιμοποιούνται τα 700 MHz για την χερσαία ψηφιακή τηλεόραση ενώ σε άλλες κατά κύριο λόγο αυτό το εύρος φάσματος χρησιμοποιείται για τη χερσαία ψηφιακή τηλεόραση. Τώρα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρε αυτές. Μα θα πρέπει εκείνες να αποφασίσουν. Αυτή η αξία για το φάσμα άνω των 700 MHz στις τηλεπικοινωνίες είναι περίπου 11 δισεκατομμύρια το χρόνο. Χρήματα τα οποία θα μπουν στον εθνικό προπολογισμό. Και από εκεί και πέρα τα κράτη-μέλη τα ίδια θα αποφασίσουν πώς θα τα αξιοποιήσουν. μπορεί να αποφασίσουν να δώσουν αυξήσεις σε αστυνομικούς και, και καθηγητές και δασκάλους. Μπορεί να θελήσουν να βοηθήσουν τους ε, παραδοσιακούς τηλεοπτικούς σταθμού. Αλλά όλα αυτά βέβαια θα έχουν κάποια όρια από, την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Πάντως θα είναι στο, κράτη, στο, χέρι, στο χέρι του κράτους μέλους να αποφασίσει Εάν κάποιο αντιμετωπίζει δυσκολίε την ώρα που θα κληθεί να ε, αλλάξει τη δραστηριότητά του από τα 700 ή άνω MHz στο ε, εύρο κάτω των 700. Και τα κράτη-μέλη από ό,τι βλέπω σε ορισμένε περιπτώσεις ε, είναι διτεθειμένα να βοηθήσουν. Περιφε... Ήπεθρος ΑΜΕΙΔΗ. Και δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη προσοχή η περισσή προσοχή στη λεπτομέρεια. Πιστεύω ότι η τυποποίηση στο βαθμό που ασχολείται με λεπτομέρειες έχει τη σημασία του εάν μπορούμε να φτάσουμε στο ίδιο σημείο για να συναντηθούμε. Αυτό σημαίνει τυποποίηση, αυτό σημαίνει πρότυπα. Θα είναι δύσκολο να ονειρευόμαστε την ε, διαλειτουργικότητα. Έγινε λόγος για ψηφιακή ταυτότητα. Πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένα πρότυπα εάν δεν είμαστε έτοιμοι να επικοινωνήσουμε και να έχουμε μια αμοιβαία αναγνώριση. Ψηφιακές ταυτότητες, ναι. Ναι, και το ξαναλέω. Ήδη έχουμε αυτό τον κανονισμό, είναι έτοιμο ο κανονισμό σύντας, αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι τομεί όπου δεν έχουν προχωρήσει τα πρότυπα αυτά. Αυτά και σας ευχαριστώ. And minutes before uh, deadline. You see? Ωραία. Ίσα ίσα φτάσαμε στην ώρα μας. Ναι, να συνεχίσω αν θέλετε, λέει ο κ. Αντιπρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε στενή επαφή και συνεργασία, να ανταλλάσσουμε απόψεις μαζί σας, κύριε Αντιπρόεδρε, για αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα της ψηφιακής ενίας αγοράς. Και άλλωστε μην λησμονούμε ότι το Κοινοβούλιο θα κληθεί να συζητήσει και τα επόμενα νομοθετήματα. επομένω μα ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μα. Κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο στι 10 η συνεδρίαση πλην των συντονιστών οι οποίοι παρακαλούνται να είναι εδώ στι 9. Στις 10 θα ξεκινήσουμε με ψηφοφορίες. Μην λησμονήσετε να φέρετε τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ εγώ που με καλέσατε. Βεβαίως εμείς θέλουμε πάντα, λέει ο κύριος Άντρους Άνσιπ, να έχουμε επαφή μαζί σας και θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε να σας ενημερώνουμε. Ευχαριστώ. Very good.